Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Έχουμε το σημείο 11, την ακρόαση για τις ε, τεχνολογίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι αλλάζει ο κλάδος. Το θέμα είναι βεβαίω πόσο βαθιές θα είναι αυτές οι αλλαγές. Και υπάρχουν πολλές συζητήσεις γύρω από το θέμα. Οι παραδοσιακές ε, οντότητες ε, βλέπουν την υπόθεση με τον νέο τρόπο, ενώ άλλες με άλλον τρόπο. Και βεβαίω εδώ στο Κοινοβούλιο, μετά από μια πρωτοβουλία της Άλντε, αποφασίσαμε να συντάξουμε μια έκθεση ιδία πρωτοβουλία για το θέμα. είναι και ο συγητής εδώ. Ε, δεν θα μακρηγορήσω βεβαίω. Θα τα δούμε μετά τα συμπεράσματα, αλλά πρέπει να είμαστε ευγνώμονε για το ότι έχουμε εδώ πέρα 7 έξοχους ομιλητέ και θα μα πούν πώ βλέπουν αυτοί το θέμα. Νομίζω πως έχουμε μερικούς πολύ καλούς ανθρώπους. Ένα θέμα πολύ επίκαιρο επίσης. Μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Υπάρχουν δύο πανέλ, όπως ξέρετε. Έχουμε χωρίσει την ακρόαση σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τις τεχνολογικές καινοτομίες και το άλλο φορά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις. Να σας συστήσω λοιπόν τους ομιλητές μας. Πρώτα απ' όλα, η Κλέρ Καρμιτζάνη, Διευθύντρια Κοινοτομίας στην Lloyds. Έχετε τον λόγο. Πέντε λεπτά θα έλεγα λίγο πολύ για να ακούσουμε και τους τέσσερις ομιλητές και μετά να ακούσουμε και τις ε, πολιτικές ομάδες και τους ε, βουλευτές. Παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ. Ευθύνεται και ένας κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας ε, κλάδος ο οποίος ε, ένα μέρος το οποίο αναπτύσσεται πάρα πολύ καλά είχε δύο επιτυχημένες τέτοιες εταιρείε, ε, την TransferWise και την Funding Cycle που έχουν φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο ο κόσμος λοιπόν αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και η αγορά φαίνεται καταποκρίνεται σε αυτήν την αγορά ο Όμιλος Lloyds παίζει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη θα επενδύσουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουμε τις ανάγκες των 28 εκατομμυρίων πελατών μας 8 εκατομμύρια εκ των οποίων ε, εξυπηρετούνται μέσω κινητών. Και βεβαίως ε, έχουμε μία σειρά προϊόντων τα οποία προσφέρουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Οπότε έχουμε κάποιους επιταχυντές αυτής της τεχνολογίας που στηρίζουν τις νέες εταιρείες ε, με επιχειρηματικό κεφάλαιο. Συνεργαζόμαστε και χορηγούμε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις ε, και έχουμε και διάφορους μέντορες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως χρονίζουμε ακόμα πως υπάρχει σοβαρή ανάγκη για να υπάρχει μια εμπειρία η οποία θα αγκαλιάζει όλους τους πελάτες μας. Υπάρχουν ακόμα 5 εκατομμύρια άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τους το διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε λοιπόν κάποια μοντέλα τα οποία είναι πάρα πολύ βασισμένα στο διαδίκτυο και ε, απαιτούν ελάχιστα κεφάλαια. Αυτό είναι πράγμα τους χάρη προφανές με πλατφόρμες όπως το Airbnb, Alibaba και Facebook. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στις 15.000 νέες εταιρείες ε, στον τομέα του FinTech, της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας ε, και βεβαίως είναι η δική μας ευθύνη να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και την προστασία των πελετών. Και πάνω να σου πω ότι έχουμε έξι πράγματα που πρέπει να έχουμε κατά νου. Πρώτα απ' όλα να υπάρχουν κάποιε παγκόσμιες προδιαγραφές ε, για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, να εναργωνιστούν οι κανόνες ε, σε, ολο... σε διάφορες χώρες και να υπάρχει φορητότητα των λύσεων. Θεωρώ πως αυτά θα βοηθήσουν ε, και την ανάπτυξη της νέα ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Το επόμενο θέμα είναι να απτυχθεί μια κουλτούρα πειραματισμού, κατά το οποίο βλέπουμε παραδείγματος χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Λόιτ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ίσο πεδίο ανταγωνισμού. Και βέβαια ακριβώς σκοπεύουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι θα πρέπει να υπάρχουν Ε, εγκαίρω δοκιμέ για να δούμε το τι γίνεται με την ιδιωτική ζωή των πελατών. Παραδείγματο χάρη στο διαδίκτυο μπορεί να υπάρχει ένα κουμπί το οποίο θα πρέπει να πατήσει κάποιο για να αποδεχτεί τα κούκκι, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι πάρα πολύ πρακτικό σε μια οθόνη κινητού. Το επόμενο θα είναι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους μηχανισμούς ε, οι οποίοι θα ανοιχνεύουν ακριβώς αυτά τα στήματα, τα οποία διαταράσσουν τις παρασυριακές δομές για να δούμε ποιοι Ακριβώς είναι οι συστημικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από κάτι τέτοιο και θα πρέπει ακριβώς να δούμε τα θέματα της κυβερνοασφάλειας ε, των δεδομένων, του διαδικτύου των πραγμάτων ε, και του νέφους. Ε. Το επόμενο αφορά την πρόθεση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων δρόντων και τη δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή. Οι οργανισμοί εστιάζουν προς το εσωτερικό τους, αλλά καθώς στρέφονται προς τα έξω θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας και θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ε, πτυχές ε, του φάσματος. Και τέλος η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική και ελκυστική σε σχέση με την Ασία και ιδιαίτερα την Κίνα και τις ΙΠΑ ε, όπου υπάρχει βεβαίως πάρα πολύ μεγάλος αγώνας για να προσελκύσουν το κεφάλαιο το επιχειρηματικό. Έτσι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις και να υπάρχει πρόσβαση σε παγκόσμια ταλέντα. Να σας πω πράγματα τώρα τα οποία έμαθα κατά τη διάρκεια της αντιδρομής μου. Το πρώτο είναι ότι σκοπεύουμε να μην αφήσουμε κανέναν θα έλεγα εγκαταλειμμένος ε, ήδη έχουμε ενισχύσει 20.000 επιχειρήσεις δεύτερον είναι να στην διάφορες προκλήσεις όπως καθόλου για να στηρίξουμε τον κλάδο και να ακούγονται οι φωνές των ε, πελατών όπως ε, παραδείγματος χάρη έκανε πρόσφατα η υποπτική αρχή της Σιγκαπούρης ε, Επίση πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη του κλάδου όχι μόνο με κεφάλαιο αλλά με αυτό το οποίο λέμε εναλλακτική χρηματοδότηση που συμπληρώνει την παραδοσιακή χρηματοδότηση και ανοίγει για τις πόρτες των μεγάλων οργανισμών για να υποστηρίξουμε την αλλαγή και βεβαίω θα πρέπει να υπάρχουν και περισσότερες γυναίκες στο ψηφιακό κλάδο. 51% των πελατών μας είναι γυναίκες. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε κάνει μια δημόσια δέσμευση για προώθηση γυναικών σε υψηλόβαθμες ε, θέσεις για να προωθήσουμε ακριβώς περισσότερες γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι μόλις 10% των ιδρυτών τέτοιων εταιριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά και αναμένουμε περισσότερο διάλογο με τον κλάδο καθώς το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν σκύβουν πάνω από το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Μάρκο που είναι ε, ε ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής ε, της ε, εταιρείας. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ε, ίσως δεν ανταποκρίνομαι στην ε, εικόνα που έχετε για τον χαρακτηριστικό ιδρυτή ε, FinTech που συνήθως είναι νέος και φοράει σχισμένο τζιν. Εγώ έχω άσπρα μαλλιά και φοράω και γραβάτα καμιά φορά, τώρα δεν έχω μαζί μου. Ε, φαίνεται ότι ο κλάδος του FinTech έχει ενηλικιωθεί, έχει σοβαρευτεί και γι' αυτό χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα σε σας. Είμαι ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας Crossings και FinTech από τη Γερμανία για Supply Chain Finance. Ε, ε, έχω όμως και μακρά εμπειρία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ήμουνα ε, πριν από λίγα χρόνια μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ε, είμαι και στο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο, τον αντίστοιχο ΕΣΠΑ. Έχουμε δηλαδή πολλά σημεία επαφής με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με Connecting Europe Facility, διάφορες γενικές διευθύνσεις και μεταξύ άλλων και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που συμμετείχα ε, σε μία ομάδα που ασχολείται με τέτοια θέματα όπως το σημερινό και άλλα με ενεργειακή τιμολόγηση κτλ. Γνωρίζω λοιπόν τη σημασία των ημερίδων τέτοιου τύπου. Από την άλλη θα προτιμούσα να είχα ασχοληθεί με άλλα θέματα τα τελευταία χρόνια για να ασχοληθώ και με την ανάπτυξη ε, της εταιρείας μου. Ελπίζω να μπορέσω να σας βοηθήσω και ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε και έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ε, τοποθετηθούμε. Σήμερα εκπροσωπώ την ιδρυθήσα ε, European FinTech Alliance. Είναι μια οργάνωση που η οποία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2016 για πρώτη φορά και ασχολείται αποκλειστικά με τεχνολογία τη χρηματοπιστωτική fintech, όχι μόνο ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διεθνώς. Ε, προερχόμαστε από διάφορους κλάδους, mobile banking, ηλεκτρονικές πληρωμές, συναγματικές ισοτιμίες και ε, συναλλακτήρια κλπ. Και προσπαθούμε να τα ενώσουμε όσο γίνεται περισσότερο όλα αυτά. Και φυσικά, ακούσαμε και προηγουμένως ότι εκπροσωπούμε ε, τον κλάδο και θέλουμε να δώσουμε φιλικές λύσεις και στις εταιρείες και στους καταναλωτές. Γιατί ε, το θέμα δεν είναι μόνο B2C, δηλαδή από επιχειρήσεις σε καταναλωτές, αλλά και B2B από επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις που θέλουν νέες τεχνολογίες. Και όλο και περισσότερο το βλέπουμε αυτό. Ε, τα θέματα αυτά είναι αλληλένδετα ε, τα τιμολόγια, οι πληρωμές, η χρηματοδότηση, η συλλογή πόρων ε, εντάσσονται στη νέα ψηφιακή εποχή και υποδομή που από εκεί θα αναπτυχθεί η οικονομία και θα δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη φυσικά. Εμείς οι Crossings αρχίσαμε με τέσσερις εργαζομένους και τώρα είμαστε πάνω από δηλαδή ε, πολύ ε, μεγάλες και ραγδαίες εξελίξεις. Αυτό δεν αφορά τον ίδιο τον κλάδο της FinTech, αλλά και τη συνεργασία ε, με άλλες δομές και με τράπεζες. Δηλαδή δεν είναι ξεχωριστός κόσμος. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παραδοσιακού τύπου. Μερικά παραδείγματα θα μπορούσα να σας δώσω χρηματοδότηση και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ έχουμε πολύ νέες δυνατότητες, νέες τεχνολογίες, ε, πέρα και από συνδεδεμένη από ε, το, την, ε, τον έλεγχο της υγείας μιας επιχείρησης, της πιστοληπτικής ικανότητας κτλ και της εξοπιστίας. Ακόμα δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες για το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και καλό είναι να ασχολούμαστε με αυτά τα νέα θέματα, να τα δοκιμάσουμε και σε συνεννόηση πάντα με τα αρμόδια όργανα να τα λύνουμε. Από την άλλη, παίζει ρόλο και σημαντικό και πρωταγωνιστικό η προστασία των καταναλωτών. Ε, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για λύσεις ε, ε, χρηματοπιστωτικής ε, τεχνολογίας, αλλά αυτές οι εταιρείες είναι πάντα νεοφυείς, δεν έχουν την παραδοσιακή ασφάλεια και βεβαιότητα που, που, και εμπιστοσύνη που εμπνέουν οι τράπεζες, αλλά έχουν την υποχρέωση να παρέχουν κάποια προϊόντα στους καταναλωτές και να τους εξασφαλίζουν. Από την άλλη, κανόνες που θα ρυθμίσουν όλο αυτό το κλάδο δεν θα πρέπει να τον στραγγαλίσουν. Γι' αυτό ε, είμαστε στη διάθεσή σας να βρούμε από κοινού ε, κάποιες λύσεις και κάποιες ρυθμίσεις. Έτσι ώστε και οι νέες τεχνολογίες να χρησιμοποιούνται και οι εταιρείε να εξοικειώνονται και να αναπτύσσεται και ο κλάδος χρειαστεί μια ρύθμιση σταδιακή και βαθμιαία ανάλογα με το ρίσκο, με τον κίνδυνο, με τις υποσχέσεις, με τις δραστηριότητες ε, που ε, είναι στην υπηρεσία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Ε, θα ακούσουμε και άλλα παραδείγματα για το PS2 αλλά και άλλα πρότυπα εναλλακτικής χρηματοδότησης και δανειοδότησης. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε πανευρωπαϊκά μια εναρμονισμένη ρύθμιση και νομοθεσία έτσι ώστε οι εταιρείε να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μια εσωτερική ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστώ πολύ Μάρκους. Και τώρα έχει το λόγο η Τάνια Κλάερ από το ε, Core Product Team Κλάρνα. Ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέψατε να έρθω σήμερα εδώ και να σας απευθύνω το λόγο. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας μην ξεχνάμε ε, ότι προσπαθούμε να επιτύχουμε καινοτομία και ποιος το προσπαθεί αυτή. Όχι εσείς, η πολιτική, ούτε εγώ, η fintechs, ούτε διάφοροι άλλοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί. Αυτό ε, το ζητάει ο καταναλωτής. Οι εταιρείε οι οποίες δεν ακούνε την άποψη του καταναλωτή δεν θα επιβιώσουν, δεν θα μακροημερεύσουν. Όταν πρόκειται για επιγραμμικές ε, πληρωμές, η εταιρεία μας ε, ε, καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη. Εμείς φτιάχνουμε προϊόντα για να είναι εύκολο να ψωνίσει κανείς επιγραμμικά. Ε, ο καταναλωτής είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας. Και αυτό το δείχνει και το ότι έχουμε 45 εκατομμύρια καταναλωτές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και πάνω από 65.000 ε, συγχωνεύσεις, ε, μάλλον αγορές ε, των δικών μας των υπηρεσιών. Έχουμε πάρα πολλές συναλλαγές και είμαστε ενεργοί σε 70 κράτη γενικώ. Πέρυσι μπήκαμε και στην αγορά των πολιτειών και το κατορτάσαμε με μεγάλη επιτυχία. Υποθέτω όμως ότι θα πρέπει άλλοι παίκτες ε, της FinTech να γνωρίζουν ότι εμείς λειτουργούμε ως τράπεζα ε, είμαστε δεσμευμένοι από όλα αυτά που αφορούν τις τράπεζες, μεταξύ αυτών και το τραπεζικό απόρριτο. Βέβαια, οι τράπεζες ε, εμποδίζουν την κινητικότητα στην αγορά, μη δίδουν στοιχεία για τους καταναλωτές και δημιουργούν σκόπιμα της τις ανεπάρκειες, τις αδυναμίες, ε, επιβάλλουν υψηλά, υψηλό τίμημα, τέλη για τις συναλλαγές. Αυτό όμως ευτυχώς αλλάζουν. Κάποια στιγμή η οικονομία της αγοράς είναι εκείνη που λέει ότι θα πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες του καταναλωτή για να είναι κανείς επιτυχημένος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει λοιπόν να άρει τα εμπόδια θα πρέπει να διασφαλίζουμε ισότιμο ανταγωνισμό και ευκαιρίες. Πρέπει να έχουμε στόχο να προστατεύουμε τους καταναλωτές μειώνοντας το κόστος των συναλλαγών. Και αν τα κάνει κανείς όλα αυτά, αυτό συμβάλλει σε μια αποτελεσματική αγορά. Εάν λοιπόν στρέψουμε το βλέμμα πίσω πριν από 10 χρόνια, τότε δεν είχαμε τα FE τηλέφωνα, ούτε τα apps, ούτε το ίντερνετ όπως τα χρησιμοποιούμε σήμερα. Τώρα όλα αυτά έχουν μπει στη ζωή μας. Η τεχνολογία ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή και ο χρηματοπιστωτικός χώρος είναι ένας από τους πιο δύσκολους τομείς όπου λαμβάνουν χώρα και ανατομίες. Επίσης, ε, όλα αυτά είναι επίμαχα γιατί οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι οι fintechs ε, τους τρώνε το ψωμί τους. Όμως τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες ε, δεν ε, κάλυψαν τις ανάγκες. Υπάρχει λοιπόν, ε, υπάρχουν λήψεις ε, και οι τράπεζες φαίνεται να έχουν ξεχάσει ποιοι είναι οι πελάτες, έπαψαν πια να αναπτύσσουν προϊόντα για τις ανάγκες τους. Κάποιοι το συνειδητοποίησαν και άρχισαν να δημιουργούν προϊόντα για τους πελάτες, πραγματικά καλά προϊόντα. Αν λοιπόν στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον, μετά από 10 χρόνια, σήμερα οι νέοι που έχουν ε, όλα αυτά τα εξυπνά, τα εφή, τηλέφωνα και πολλά άλλα, αυτοί ε, θα θέλουν να κάνουν, τα, να χειρίζονται οικονομικά τους ε, εξίσου με τρόπο, δεν θα καταφύγουν στις παραδοσιακές τράπεζες. Οι καταναλωτές αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και γι' αυτό νέες υπηρεσίες, νέες επιχειρήσεις αρχίζουν να προσφέρουν ευπρόσδεκτες υπηρεσίες. Αυτό αφορά και τις τράπεζες. Και εμείς ως εταιρεία FinTech καλωσορίζουμε τον ανταγωνισμό. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν οι νομοθέτες και οι πολιτικοί να συμβάλλουν σε αυτή την αλλαγή, μπορούν να το κάνουν δίνοντας δυνατότητα στους καταναλωτές να ε, κινητοποιήσουν την ε, ε, νομοθεσία. Έχουμε σαφείς προδιαγραφές, αλλά αυτές σκοτώνουν την καινοτομία. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα μια μηχανή ε, με πολλές λεπτομέρειες, πώς πρέπει να είναι αυτή η μηχανή. Αν υπάρχουν όμως ε, τόσες πολλές λεπτομέρειες, κανείς δεν θα κάνει δοκιμές. Το ίδιο και για έναν regulator στην FinTech. Θα καταλήξουμε τελικά σε ένα πλαίσιο που δεν θα είναι συμβατό με την καινοτομία και μόνο αυτό δεν θα είναι συμβατό και με αυτά που επιτιμεί ο καταναλωτής. Τελειώνοντας λοιπόν, ε, απευθυνόμαστε σε εσά ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εκδώσετε νομοθετικές πράξεις που θα βοηθήσουν ε, να προστατεύονται οι καταναλωτές ε, και όχι οι κύριοι πάροχοι, οι παραδοσιακοί πάροχοι. Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιες αρχές να κάνουν την εποπτεία και όχι η παραδοσιακοί πάροχοι. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει κανείς τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που επιθυμεί και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με ασφαλή τρόπο. Οι νομοθέτες ε, θα πρέπει να εξάρουν περισσότερο την απόδοση και όχι τις λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές. Και η νομοθεσία δεν σημαίνει ότι δεν προστατεύεται ο καταναλωτής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο τελευταίο σε Ερτερνάς που είναι πρόεδρος. <clears throat> Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή σας που προσκάλεσε την ΥΠΑΛ να κάνει κάποια σχόλια. Θα πω λίγα λόγια για τις συνεργασίες που έχουμε μεταξύ των εφισταμένων και των παλαιών δρόντων στην FinTech και κάποια από τα ζητήματα για τις ρυθμιστικές αρχές. Νομίζω πως θα έλεγα αυτός ο γάμος τεχνολογίας και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν είναι κάτι το καινούριο. Ξέρετε, πάντα οι υπηρεσίες αυτές ε, ε, άλλαζαν με την τεχνολογία. Αν δούμε τις πλαστικές κάρτες, ε, τα μηχανήματα αναλήψεων. Βλέπουμε όμως τώρα τη δυνατότητα μιας επιτάχυνσης ε, των εξελίξεων, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, γιατί μιλάμε πλέον για μια παγκόσμια διάδοση και του διαδικτύου και των έξυπνων τηλεφώνων. Σε σχέση με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για να σκεφτούμε με πράγματα, υπάρχουν βεβαίω πολλέ προκλήσει. Πολλέ εταιρείε χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να ξανασκεφτούν εντελώ ε, πώ παρουσιάζονται οι φυστάμενε υπηρεσίε. Και νομίζω πως ε, θα έχουμε πολλέ και συναρπαστικέ εξελίξει που θα προκύψουν από το πώς οι εταιρείε αυτές είτε συνεργάζονται με τα υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά. Είτε δηλαδή είναι ένα επιπλέον στρώμα, είτε είναι συνεργασία για συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να ενδυναμώσουν κάποιες υπηρεσίες ε, για να τις κάνουν πιο αποτελεσματικές και φτηνές. Ε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, παρά το ότι ε, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα είναι κάπως αργά και δεν ακριβώ τα καταφέρνουν τόσο γρήγορα να διατηρήσουν πελάτες για πολλές εταιρείες fintech προσπαθούν να λύσουν ένα συγκεκριμένο ζήτημα ε, και ίσως να μην θέλουν να γίνουν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα απλά τους ενδιαφέρει ακριβώς η κλίμακα ε, το ότι έχουν έτσι ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό θα έλεγα και ως PayPal εμείς είμαστε μια εταιρεία 18 ετών, ε, ήμασταν πάντα μια εταιρεία fintech. Αυτό το οποίο καταφέραμε ήταν να γίνουν ε, τέλειες θα έλεγα χωρίς καμία τριβή ή ψηφιακές πληρωμές ε, έτσι ώστε για τους εμπόρους να μην έχει σημασία το πώς ήθελε να πληρώσει ο, ο και για, την πλευρά του καναλτή το ότι ήμασταν κατοβολικό και έμπιστο Πέρυσι επεξεργαστήκαμε 5 δισεκατομμύρια πληρωμές, έχουμε 192 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίω. οπότε υπάρχει κλίμακα στις αγορές αυτές. Είναι αγορές μεγάλης κλίμακας. Τώρα υπάρχουν κάποια ρυθμιστικά ζητήματα. Όταν μιλάμε για fintech είναι κάπως παραπλανητικό ε, το θέμα, γιατί δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Αυτό το οποίο βλέπουμε Και βεβαίω υπήρχε και πριν από 15 μέρες ε, ε, βλέπουμε Είχαμε ένα συνέδριο που βλέπουμε Σιγκαπούρη, Λονδίνο και άλλα παραδοσιακά θα έλεγα χρηματοπιστωτικά κέντρα που προσπαθούν να διατηρήσουν τον ρόλο του και άλλε χώρε στην Νοτιοανατολική Ασία που χρησιμοποιούν τη φινιτεκ ακριβώ για να περιλάβουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, αναψώμενες οικονομίε όπω η Ινδία που προσπαθούν έτσι να έχουν μια μεγαλύτερη εποπτεία και να αναπτύξουν και μια οικονομία χωρί μετρητά η οποία θα είναι καλύτερη για πολλού και διάφορου λόγου. Και όπω είπαν και οι συνάδελφοι, ακριβώς ε, υπάρχει αυτή η ιδέα του ε, χώρου πειραματισμού γιατί ό,τι και αν προκύψει από εκεί ένα από τα σημαντικότερα και ευχάριστα ζητήματα είναι πως ε, θα μπορέσουν έτσι να έρθουν σε επαφή ρυθμιστικές αρχές και αυτοί οι οποίοι καινοτομούν και έτσι δεν θα υπάρχει πια φόβος ε, εκατέρωθεν. Οπότε ό,τι και να συμβεί νομίζω θα είναι θετικό. Υπάρχουν τρία ζητήματα τα οποία θα έλεγα εγώ ότι χρειάζεται για να προωθηθεί υπεραιτέρω το Κάποια από αυτά αναφέρθηκαν ήδη. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτών των υπηρεσιών ε, υπάρχουν απαιτήσει που λέγονται know your customer ε, για να ξέρουμε ποιοι είναι οι πελάτες μας σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος. Αυτό πρέπει να γίνει σωστά Αλλιώς ε, θα καταλήξουμε με αναποτελεσματικά μέτρα ε, τα οποία θα επαναλαμβάνονται συνεχώς. Πρέπει παραδείγματος χάρη η τηλεταυτοποίηση να είναι εφικτή για τέτοιες εταιρείες για να, είναι, για να είμαστε επιτυχημένοι. Κατόπιν για την ασφάλεια. Οι συνάδελφοι το ανέφεραν ήδη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενθαρρύνω να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιες υπηρεσίες ταυτοποίησης ε, που θα βασίζονται στον κίνδυνο, σε ένα προφίλ κινδύνου. Και τέλος να μπορούν οι υπηρεσίες στην Ευρώπη να έχουν ένα διαβατήριο, όπως το λέμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανέφεραν οι συνάδελφοι ότι δεν είναι ακόμα εφικτό λόγω του κατακρεματισμένου ρυθμιστικού πλαισίου. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Θα σταματήσω εδώ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε και ευχαριστώ να ακούσουμε για την έκθεσή σας αυτή που είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ επιτυχημένη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν το πρώτο γύρο ε, των προσκεκλημένων μας και τους ευχαριστώ που ήρθαν. Τώρα έχουμε ένα γύρο ε, των Ευρωβουλευτών τα μέλη της Επιτροπής μας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια της έκθεσης αυτής, που είναι η κυρία Κόρα Βανιουενχόιζεν. Δεν ξέρω αν το είπα και πώς βγήκε η Κόρα. Thank you, Mr. Chairman. That's the reason why most people just call me Cora. Γι' αυτό με λένε η Κόρα οι περισσότεροι. Τώρα καταλάβατε γιατί. <laughs> Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που ήρθαν σήμερα στις Βρυξέλλες να μας μιλήσουν. Εγώ ανέλαβα την πρωτοβουλία φυσικά να καταθέσω ένα σχέδιο έκθεσης για τα προϊόντα FinTech, γιατί οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται με τέτοιο ραχδαίο ρυθμό και ταυτόχρονα όλες, που θέλουμε στην Ευρώπη να έχουμε και εμείς το μερίδιό μας ε, στην παγκόσμια πίτα της οικονομίας, για να το πω έτσι. Εσείς αναφερθήκατε πάρα πολύ ε, σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα που συνδέονται με το FinTech, αλλά τι πιστεύετε ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να εθαρρύνουμε την καινοτομία ε, στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε ε, στον κατακαιρματισμό της νομοθεσίας και στην πολλή διάσπαση και θέλετε μεγαλύτερη εναρμόνιση από ό,τι ακούω δεδομένων των προαπαιτουμένων για την προστασία των καταναλωτών από τη μια και την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την άλλη. Πώς πιστεύετε ότι οι νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν περισσότερο την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να έρθουμε πιο γρήγορα στην Ένωση Κεφαλαίου Αγορών που όλοι επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κόρα. Λοιπόν, Ακολουθούν οι σκιώδεις αν θέλουν να μιλήσουν. Ε, ο κύριος Χένς. Thank you very much indeed, uh, President. Um, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπε και η κόρα, θέλω και εγώ να καλωσορίσω ε, όλους τους ομιλητές μας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και εκτιμώ πολύ την παρουσία σας. Και όπως είπε και η κόρα, παλεύουμε με αυτό το ζήτημα και Δράτω με τις ευκαιρίες των όσων είπε κύριος Νάς για την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών και τι επίκειται ως προς ζητήματα ασφαλείας. Ε, παρακολουθώ όλα αυτά που λέτε και τις παρατηρήσεις σας. Εσείς αναφέρεστε στην υφιστάμενη νομοθεσία. Αυτή θέλετε να ε, αλλάξει λόγω των ε, μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών. Θέλετε να, να προσαρμοστεί η παλιά νομοθεσία ή χρειάζεται να αρχίσουμε από μηδενική βάση. Αυτό ερωτώ. Είναι αρκετή νομοθεσία για να μπορέσει να τροποποιηθεί και να ενημερωθεί, ε, ας πούμε, ή χρειάζεστε από την αρχή η χρειάζεται απο την νομοθεσία. Τάνια ταγια μιλησε για ε, τη ζήτηση των καταναλωτών που αυτοί οθούν για να γίνουν αλλαγές σε αυτό τον κλάδο και μάλιστα έγιναν και πάρα πολύ γρήγορα και έχετε απολύτω δίκιο. Αλλά εγώ ρωτώ για την νομοθεσία την ίδια. Εδώ μιλάμε για ε, αναρρύθμιτες ε, λειτουργίες και δραστηριότητες. Έχουν όλοι τη δυνατότητα να λύνουν τα προβλήματα ε, με τρόπο πρακτικό, έχουν την ε, τεχνογνωσία δηλαδή και τη δυνατότητα. Η FCA που γνωρίζω εγώ έχει βάλει στην εντολή της ε, και αυτό το στοιχείο ανάπτυξη τεχνολογίας έτσι ώστε να φτάσουν σε σημαντικούς στόχους. Ε, άλλες ρυθμιστικές αρχές δεν ακολουθούν αυτό το στόχο. Εσείς πώς το βλέπετε αν είναι καλή η νομοθεσία και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου και των καταναλωτών κυρίως. Αυτό τι σημαίνει. Ε, χρειάζεται νέα νομοθεσία ή απλώς προσαρμογή της παλιάς. Θα παρακαλούσα να μου απαντήσει. Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Ότι εντάξει και οι νομοθέτες μαθαίνουμε, αλλά θυμηθείτε τι είχε γίνει, ένα τεράστιο κράχ ε, σε κάποια κράτη-μέλη, όπου οι τράπεζες δεν ε, είχαν τον τρόπο ούτε τα μοντέλα να κατανοούν τον κίνδυνο. Και θα ήθελα να ρωτήσω αυτά τα νέα προϊόντα μπορούν να βοηθήσουν τον τραπεζικό τομέα να εκτιμήσουν τον κίνδυνο. Γιατί αυτό είναι μία από τις κύριες δουλειές της τράπεζας, να καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Αλλιώς δεν μπορεί να δανείζει χρήματα μια τράπεζα και να δουλεύει πραγματική οικονομία. Μπορεί να τους βοηθήσει η fintech να κατανοήσουν πώς θα διαχειρίζονται το κίνδυνο μεγάλες και μικρότερες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστές, η κυρία Μπερέ. Ευχαριστώ. Και πάλι με ο Κατελίν Ιβάν, γιατί έχουν προεκλογική εκστρατεία στη Ρουμανία. Ευχαριστώ. Μπαίνουμε τώρα σε ένα έδαφος που η Ευρώπη θα πρέπει να είναι στην αιχμή της καινοτομίας και να μην τη φρενάρει αλλά να μην καούν και τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Θα πρέπει οι σχέσεις fintech και τραπεζών να βασίζονται σε μια καλή συνεργασία, έτσι, με εταιρική σχέση. Και εσείς τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για να επιτύχει αυτή η εταιρική σχέση. Εσείς είστε εμπειρογνώμονες όλοι σε αυτόν τον κλάδο. Πώς το βλέπετε. Πώς αναλύεται τις αδυναμίες ή και τις ε, δυνατές ε, πτυχές της ευρωπαϊκής αγοράς σε σύγκριση με την αμερικανική. Επόμενη ερώτηση. Και ελπίζω να έχετε το χρόνο να απαντήσετε σε όλα αυτά. Εσείς πώς ε, βλέπετε τους συγκεκριμένους κινδύνους σε ό,τι αφορά τις πληρωμές και μιλώ για την ασφάλεια των πληρωμών και την καταπολέμηση της απάτης. Και μη μας πείτε, εντάξει, η φυσική απάντηση θα ήταν αφήστε μας να αναπτυχθούμε γιατί αλλιώς φρενάρετε την καινοτομία και μετά θα είναι πολύ αργά όταν έρθουν πολλαπλές οι απάτες. Τι προτείνετε εσείς για να μπει ένα φρένο στην απάτη από την αρχή. Και μετά για το τραπεζικό μοντέλο. Έχω διπλή ερώτηση. Πρώτον, τι πιστεύετε ως προς τον αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας στις τράπεζες. Δηλαδή, θα υπάρξει επανάσταση, εντάξει θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά χάνονται και άλλες. Το έχετε μελετήσει, έχετε καμιά ιδέα για την τάξη μεγέθους και για το επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών. Πιστεύετε ότι η διαχείριση κινδύνου που συνδέεται με το FinTech ε, αμφισβητεί τα εσωτερικά μοντέλα λειτουργίας σε πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες. Ευχαριστώ ε, κυρία Μπερές. Από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης και τους ε, προσκεκλημένους μας ε, για τις ομιλίες τους. Ελέγχθη ότι FinTech αφαιρεί την ένταση από το σύστημα και καθαρά οικονομικά το κόστος ε, συναλλαγής έχει μειωθεί πάρα πολύ και θα μειωθεί περαιτέρω και στο μέλλον. Και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι οι αγορές γίνονται πιο αποτελεσματικές και αυτό πρέπει να το στηρίξουμε με νομοθεσία. Κατά την άποψή μου όμως αυτό έχει το μειονέκτημα ότι οποτεδήποτε προκύπτουν αστάθειες, οι αστάθειες αυτές ε, ε, εξελίσσονται πολύ πιο εύκολα κλιμακώνονται πολύ πιο εύκολα. Παραδείγματο χάρη ισχύει το εξή. Υπάρχουν κάποιε μελέτε που δείχνουν ότι με την ε, εξέλιξη FinTech οι παραδοσιακέ ε, τράπεζε ε, θα μπορούσαν να χάσουν μέχρι και 40% από το τζίρο που έχουν με τον τελικό καταναλωτή. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει το εξή. Τελικά, αν υπάρξει τέτοια μεγάλη μετατόπιση στον τομέα του τελικού χρήστη είναι τόσο μεγάλο το περιθώριο, ε, θα πρέπει να σκεφτούμε σε περίοδους κρίσης ε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι είδους ε, τροχοπέδες μπορούμε να εντάξουμε έτσι ώστε να μπορούμε γρήγορα να κατευθύνουμε την αγορά οι κρατικές παρεμβάσεις πάντα είναι αργότερες και εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν να γνωρίζω ο κλάδος τι έχει να προσφέρει έτσι ώστε να μπορούμε να επέμβουμε εμείς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ακόμα και πριν επέμβει ε, το κράτος. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Φωστόχα, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά την Κλάρνα, την Τάνια Κέρν. Και θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Η καινοτομία είναι ε, μια διαδικασία που δεν μπορεί να προβλεφθεί. Έχει λεχθεί ότι είναι ο ανταγωνισμός ως μια διαδικασία εφευρέσεων. Η καινοτομία οδηγεί σε καλύτερη κατανομή των ε, προϊόντων το θέμα είναι ότι ένας κεντρικός φορέας ε, δεν μπορεί να προγραμματίζει καλύτερα και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν γνωρίζουμε ποια θα ήταν η καλύτερη λύση. Η συνέργεια των δυνάμεων είναι εκείνη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες λύσεις και τελικά να προκύψει κάτι το πραγματικά καλύτερο. Άρα δηλαδή ο ανταγωνισμός όπως σας τον περιέγραψα σημαίνει ότι έχει νόημα να περιοριστεί η διαδικασία του ανταγωνισμού, να τον βάλει κανείς ε, μέσα σε κάποια όρια και εμείς ε, στο Κοινοβούλιο αυτό που κάνουμε δεν είναι άραγε μείωση των καινοτόμων δυνατοτήτων των εταιριών FinTech. Για να το ρωτήσω αλλιώς, τι είναι εκείνο που οθεί την καινοτομία και τι πρέπει να κάνουμε εμείς στο Κοινοβούλιο για να μην σας βάζουμε τροχοπέδες και για να αφήνουμε μεγάλο περιθώριο ε, στην καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ, Μπέτρης. Πολλές ερωτήσεις τέθησαν. Ας κάνουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσω με τη σειρά που επιθυμείτε, δεν θα σας επιβάλλω εγώ. Παρακαλώ, απαντήστε στις ερωτήσεις με τη σειρά. Η ε, ε, ε, λέτε για την καινοτομία και πώς μπορούμε να την ενθαρρύνουμε. θα πρέπει να συνεργάζονται οι δικές μας εταιρείες και οι τράπεζες. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο το σύστημα λειτουργεί πολύ καλά. ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό το θέμα, συνεργαζόμαστε και με τις τράπεζες. Καμιά φορά είναι πολύ βασική συνεργασία, καμιά φορά είναι σε συμβουλευτικό πλαίσιο με τους ε, εμπειρογνώμονες και άτυπο. Δεν είναι πάντα συγκεκριμένο. Ρωτάμε ποια είναι τα παραδείγματα, τι συμβαίνει. Um, και οι τράπεζες έχουν επιταχυντές έχουν διάφορα προγράμματα ξέρω εγώ, 20 εταιρείε σε βάση διετία ή τριετία και παρακολουθούν πώ εξελίσσεται η κατάσταση. Αυτά αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα στην Ευρώπη. Ε, τα μοντέλα λειτουργούν διαφορετικά. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ποιες είναι οι βασικές ανάγκες ε, για την νομοθεσία. Και αυτό είναι αμοιβαία εποφελές να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία πραγματικά θα παρότρινα να μην τα βλέπουμε ξεκομμένα αυτά. Και η Κλάρνα πραγματικά ε, ασχολείται με αυτά τα θέματα από την αρχή, πλησιώνει τον πελάτη από τα πρώτα στάδια ε, και οι περισσότερες εταιρείες είναι νεοφυείς, startups ε, και πραγματικά αγωνιζόμαστε έτσι να αγκαλιάσουμε, να υιοθετήσουμε τον πελάτη κυριολεκτικά. Μια ερώτηση που μου έγινε συγκεκριμένα και άμεσα, γιατί εργάζομαι 10 χρόνια σε αυτό τον κλάδο, τι έχω διαπιστώσει. Οι ε, startups ξεκινούν από πάρα πολύ μικρά σχήματα ε, και στην αρχή είχαν προβλήματα ε, για τις πληρωμές, μετά είχαν προβλήματα με τα δάνεια, αλλάζουν, δεν έχουν πάντα τα ίδια προβλήματα, μετά είχαν προβλήματα παροχής συμβουλών και τώρα προχωρούμε προς ε, ε προγράμματα ασφάλισης, insurtech, όχι fintech δηλαδή, ε, στο Ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, εταιρείε, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ασία και στην Κίνα και το fintech δεν είναι κάτι το ενιαίο και όταν κοιτάτε για την νομοθεσία θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχει οριμάσει ο καιρός ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός παρακολούθησης όχι μόνο νομοθεσία και το βασικό είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η προστασία του πελάτη υποδομές, ό,τι έχει να κάνει με προστασία των δεδομένων και αυτή η εναρμόνιση θα πρέπει να γίνει σωστά ε, σε αυτή τη νομοθετική προσπάθεια. Αυτά, δεν ξέρω αν απάντησα σε κάποιες από τις ερωτήσει, σας. Ευχαριστώ πολύ. Η Τάνια. Ευχαριστώ. Υπήρχαν κάποια ζητήματα. Το ένα ερώτημα ήταν αν υπάρχει η σημερινή νομοθεσία και επίσης το εάν οι φυτάμενες ρυθμιστικές αρχές έχουν τις γνώσεις και ικανότητες να ρυθμίσουν τον κλάδο. Η απάντησή μου είναι ναι και όχι. Η πρωτοβουλία αυτή δηλαδή ήταν ε, φανταστική προς την κατεύθυνση της FinTech γιατί επέτρεψε σε νέες υπηρεσίες και εταιρείες να δραστηριοποιηθούν και ταυτόχρονα έβαζε τους ε, καταναλωτές στο προσκήνιο και μας έδινε δυνατότητα να έχουμε ίσορους ανταγωνισμού. Η οδηγία για το πακέτο για τις, ε, με η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών. Επίσης, υπήρχε αυτή αυτό το σκεπτικό το ότι η ασφάλεια συχνά χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να παρεμποδίσουμε την καινοτομία και υπάρχει αυτός ο φόβος της καινοτομίας που οδηγεί πραγματικά στο να εμποδίζουμε την ευελιξία και την ευκολία του πελάτη και το να έχουμε μία ενιαία και αυστηρή προσέγγιση εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι ο σωστός τρόπος ρύθμισης του κλάδου και επίσης απορρίπτουμε την ιδέα ότι οι εταιρείε αυτές δεν θέλουν εποπτεία και ρύθμιση. Το θέλουν. Πρόκειται για μια παρεξήγηση και επιχειρωμένη κιόλα. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ρυθμίζονται αυτές οι εταιρείε όπως και θα ρυθμίζονται άλλωστε υπό την δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών γιατί έτσι θα έχουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα μπορούν να ανταγωνιστούν σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε κάποιες αρχές όταν νομοθετούμε. Πρέπει να διασφαλίζουμε βέβαια ότι οι καταναλωτέ θα είναι στο προσκήνιο και να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους. Θα πρέπει επίσης ε, το επίπεδο εφαρμογή 2 να συμμορφώνεται με τις αρχές ε, του GDPR και την δυνατότητα του της φορητότητας. Θα πρέπει δηλαδή να μπορεί κανείς ως καταναλωτής να παίρνει μαζί τα δεδομένα του σε όποιον πάροχο θέλει. Πρέπει να υπάρχει τεχνολογική ουδετερότητα και να μην υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος θα πριμοδοτεί κάποιες ε, τεχνολογίες. Π.χ. να πάμε προς ε, μια βάση API. Το API είναι καλό, με παρεξηγείτε, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείουμε άλλες ε, τεχνολογίες όπως το direct access και πρέπει να διασφαλίσουμε και την αναλογικότητα βεβαίως με μια εύρωστη εποπτεία. Οπότε προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρα. Α, αισθάνομαι ότι σου παίρνω το μικρόφωνο τέλος πάντων. Νομίζω ότι πολλά από αυτά τα οποία είπε η Τάνια είναι πάρα πολύ σωστά και απαντούν στις ερωτήσεις για την κουλτούρα της ε, καινοτομίας και κάποιες ερωτήσεις για το πώς οι ρυθμιστικές αρχές βλέπουν τα ζητήματα αυτά και αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπερές για το πώς θα υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας ευθύς εξ αρχής. Νομίζω ότι η FinTech θα παίξει κέριο ρόλο στην αντιμετώπιση πολλών τέτοιων ζητημάτων και καταπολέμησης της απάτης κτλ. Αυτό είναι νομίζω ένας από τους τομείς που προσελκύει περισσότερο τις εταιρείε αυτές για να αναπτύξουν τα προϊόντα τους γιατί ξέρουν ότι έχουν φοβερές ευκαιρίες να πουλήσουν το προϊόν σε όλες τις υπόλοιπες εταιρείε του κλάδου. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα ε, σε αυτό το πεδίο πολύ ενθαρρυντικά και είναι πάρα πολύ αναφέρθηκαν στο PayPal. Ε, ως ε, αναφέρθηκαν στο PayPal στην αρχή ως μια εταιρεία διαχείρισης κινδύνου. Αυτό το οποίο δηλαδή προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι θα καταλαβούμε, θα καταλαβαίνουμε πότε κάτι ήταν πολύ επικίνδυνο και το καθαίρουμε Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μια εμπιστοσύνη στην δική μας εταιρεία, όπως και σε άλλες εδώ σε αυτό το πάνελ. Νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όσον αφορά το πώς το βλέπουν οι ρυθμιστικές αρχές. Αναφέρθηκε η FCA, η Βρετανική Ρυθμιστική Αρχή, που είναι πιθανότατα η πιο πρωτοποριακή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αν αρχίσουν να έχουν ρυθμιστικές αρχές ε, τμήματα fintech είναι όπως ε, στην αρχή οι εταιρείε έχουν τμήματα e-commerce ε, και τώρα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να είναι 100% μέρος δουλειά τους, αλλιώς δεν θα επιβιώσουν. Πρέπει λοιπόν ακριβώς να επιταχυνθεί αυτή η πορεία. Θεωρώ λοιπόν πως υπάρχουν πολλοί λόγοι να είμαστε αισιόδοξοι. Οι ρυθμιστικές αρχές ανταποκρίθηκαν παγκοσμίω ε, είχαν να αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα που προέκυψαν από την τραπεζική κρίση, τον κανονισμό της βασιλείας και τι έπρεπε να κάνουν με αυτό. Αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο αισιοδοξία και μια τελευταία παρατήρηση για την Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών και Φίντεκ νομίζω. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Η ιδέα αυτή του τι μπορούν να κάνουν οι εταιρείε fintech για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς ε, τέτοιες υπηρεσίες για μισά, για μικρά ποσά σε ευρώ αλλά με τρόπο που θα προωθήσουν την ασφάλεια τότε θα ήθελα να σα ενθαρρύνω να είστε κάπως πιο ανοιχτό μυαλί σε αυτό. Έχουν γίνει πολλά θετικά πράγματα, ειδικά στη ΣΥΠΑ, που μπορούν εύκολα να γίνουν στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να υπάρχει, όπως είπαμε, δυνατότητα μεταφοράς αυτών των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, Μάρκος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εντάξει, δεν ξέρω αν κατέγραψα όλες τις ερωτήσει σωστά. Θα πω τα σημαντικότερα, κατά τη γνώμη μου. Καταρχήν, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετέ νομοθετικέ ρυθμίσει, Αν δούμε λιγάκι την ίδρυση επιχειρήσεων με τέσσερις ε, εργαζόμενους. Ε, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ε, τι είδου προποθέσει ισχύουν στην Ευρώπη για να μπορεί κανείς και να τις εφαρμόσει. Και αυτό παρεμποδίζει την ανάπτυξη μιας εταιρεία. Κατόπιν τούτου. Ίσως να οφείλεται και εκεί το γεγονός ότι είναι στενά συνδεμένα τα θέματα. Ε, τα τιμολόγια με πολλές άλλες προϋποθέσεις. Το θέμα είναι ότι ε, πράγματι υπάρχει αυτή η της σχέση. Από την άλλη βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και μία βάση για την ύπαρξη μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη. Γιατί μόνο έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα μπορούν να πηγαίνουν ε, σε μία τράπεζα για να ζητάνε χρηματοδότηση, αλλά θα μπορούν να ζητάνε χρηματοδότηση και από άλλες χώρες. Βεβαίως ε, με τα χαρτιά αυτά δεν γίνονται. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι θα πρέπει κανείς να δει λιγάκι τις ε, ισχύουσες προϋποθέσεις, να τις προσαρμόσει στους ε, ε, παρόχους γιατί είναι διαφορά το να ε, λειτουργώ ως τράπεζα ή ως μικρή επιχείρηση. Νομίζω ότι αυτός είναι σημαντικός παράγον. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο και αυτό το διαπίστωσα και στην εργασία μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ουδετερότητα της τεχνολογίας ως ε, νομοθέτες ε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πάντα τι θα κάνει η τεχνολογία μετά από 2-3 χρόνια. Άρα δηλαδή εδώ πρέπει να ισχύει ότι στην τεχνολογία ε, καταρχήν ισχύει η ουδετερότητα, τα πόσον ε, θα επικρατήσει η ηλεκτρονική υπογραφή ή όχι, αυτό θα το κρίνει ε, η αγορά. Και τελευταίο και σημαντικό, ε, πρόκειται πράγματι για την εναρμόνιση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω δει πολύ συχνά οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν ως στόχο την εναρμόνιση τελικά όμως οι διαφορές στις χώρες έγιναν ακόμα πιο έντονες από ό,τι πριν από την οδηγία. Και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να είναι ο στόχος ενός τέτοιου κανονισμού. Ειδικά αν δει κανεί ε, ότι είναι σημαντικό ε, να βρίσκεται μια αγορά σε ανταγωνισμό με την Ασία και με άλλες περιοχές όπου δεν ισχύει αυτή η περίπλοκη δομή και όπου είναι πολύ πιο εύκολο να χρηματοδοτηθεί κανείς ε, για να μπορεί και να επικρατήσει στην ευρωπαϊκή αγορά. Άρα δηλαδή θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους τέσσερις. Ε, πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε αμέσω ε, στο δεύτερο πάνελ, στη δεύτερη ενότητα. Προκλήσεις και ευκαιρίες. Έχουμε τρεις ομιλητές. Πρώτος είχε προβληθεί ο Στίβεν Μαγιόρα, δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει για λόγους απεργίας ε, και κάποια άλλα προβλήματα στη Γερμανία. Τον αντικαστά Γιάκου Μίχαλικ από την ΕΣΜΑ επίσης από το νομικό τμήμα και θα μας δώσει τις ε, δικές του απόψεις για τη ρύθμιση και την εποπτεία. Στη συνέχεια έχουμε άλλους δύο ομιλητές τον Greg Φαν Έλσεν από την BEUC και τον Τζέσι Μακουότερς από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Μέσω βίντεο διάσκεψης είναι ο τελευταίος ομιλητής μας. Ε, ήδη ε, έχει συνδεθεί και τον καλωσορίζουμε. Θα δώσουμε λοιπόν αμέσως το λόγο στον Γιάκοπ Μίχαλικ. Πέντε λεπτά θυμίζω ο καθένας ε, και μετά συζήτηση για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι βουλευτές λίγο. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για την απουσία του Προέδρου Στίβ Μαγιόρ, γιατί ματαιώθηκε η πτήση του και δεν μπόρεσε να φτάσει. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που έχει έσμα να παρευρίσκεται σε αυτή την ακρόαση. Θα σας παρουσιάσω ε, κάποιες απόψεις από τους ρυθμιστές ε, της ΕΣΠΑ ο κλάδος των fintech είναι και διατομεακός και γίνεται κοινή δουλειά ε, από, με άλλους ρυθμιστές όπως είναι η ε, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή EBA. Να αρχίσουμε μερικά γενικά σημεία. Γενικά η καινοτομία και τα προϊόντα που συζητούμε σήμερα ε, είναι ακόμα στα σπάργανα και δεν ε, ε, ε, εμποδίζουν, δεν διαταράσσουν πάρα πολύ τη λειτουργία των υφισταμένων δομών. Είναι καινοτόμα προϊόντα ανάλογα με την προσέγγιση που χρειάζεται κάθε φορά και θα πρέπει να ερευνήσουμε, να σταθμίσουμε και να εξετάσουμε για μας έχει μεγάλη σημασία η προστασία των επενδυτών και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα έχουμε υπόψη. Πολλοί ε, ρυθμιστές έχουν μια ε, ιδιαίτερα προσεκτική και συγκρατημένη προσέγγιση, ενώ οι νεοφύσιοι επιχειρήσεις θέλουν να αναπτυχθούν γρήγορα. Ε, νέες τεχνολογίες καμιά φορά χρειάζονται και δομές έτσι, διαμεσολάβησης και αρμπιτρά. Το συζητάει η Επιτροπή σας ε, στα πλαίσια του PSD2 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών. Στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ασία ο κλάδος των ε, fintech ε, προχωρεί πολύ και στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε συνεχώς σε επαφές με εθνικούς και διεθνείς ρυθμιστές για να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα ωφέλη αλλά και ποια είναι οι κίνδυνοι και ευκαιρίες ε, σε σχέση με αυτές τις εξέλιξεις. Και η IOSCO επίσης είναι μια καλή πλατφόρμα για την ανταλλαγή αυτών των απόψεων για τις εξέλιξεις. Το crowdfunding για τις ε, επενδύσεις, εμείς παρουσιάσαμε το Δεκέμβριο του 2014 ε, τις απόψεις μας και έκτοτε δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ε, χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή ρύθμιση και κάποια στοιχεία του MIFID επίσης βρίσκουν εδώ εφαρμογή. Έχουμε προτείνει κάποια ε, μέτρα, έχουν ε, προταθεί από 9 κράτη-μέλη, αλλά ε, βεβαίω υπάρχει και το θέμα των διασυνοριακών επενδύσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ έτσι, αντιφατικό σε σχέση με αυτό που προτείναμε το 2014. Παρ' όλα αυτά παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις εποπτεύουμε. Υπάρχουν 28 αρμόδιες εθνικές αρχές και εμείς διαπιστώνουμε ότι αυξάνεται και ο όγκος που ε, διακινείται. Είναι περίπου στα 525 εκατομμύρια το 2015. Σε ό,τι αφορά τώρα την αυτόματη ε, λειτουργία ε, στην ΟΝΕ, γενικότερα και στην πράσινη βίβλο για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής, το Automated ε, Advice, ε, αφορούν διάφορους πελάτες με διάφορα χαρτοφυλάκια. τώρα βρισκόμαστε και πάλι σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Στην Ευρώπη είναι λιγότερο από 1% αλλά θα αυξηθεί μέχρι το 2020 από 600% μέχρι 2.500%. Επίσης, μπορεί αυτό να συμπληρώσει ένα σύστημα παροχής συμβουλών ε, επιπληρωμή, ε, η αυτόματη παροχή συμβουλών. Στην ΕΣΜΑ έχουμε ε, γνώση και παρακολουθούμε το σύνδεσμο της αγοράς ε, με αυτούς ε, τους νέους ε, τρόπους λειτουργίας στον Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία και στην Ελβετία πρόσφατα. Το ρυθμιστικό πλαίσιο, νομοθεσία έχει να κάνει με το τα IDD, PRIPS, όλα αυτά τα αρχικά, MCD. Ε, αυτά προς το παρόν αρκούν. Μπορεί να προκύψουν και άλλοι κίνδυνοι που πρέπει να καλύπτονται. υπάρχει η κοινή η μεικτή επιτροπή ε, που θα συνεδριάσει, μάλλον θα εκδώσει την έκθεση της ε, το Δεκέμβριο. Πέρσι το Δεκέμβριο έχει συνεδριάσει. Για το DLT, από τον Απρίλιο του 2015 ε, το εξετάζουμε. Έχουμε ένα έγγραφο συζήτησης για να δούμε τι λένε οι ενδιαφερόμενοι και ο κλάδος. Και σε αρχές του 2017 θα κυκλοφορήσουν ε, οι απόψεις αυτές. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι ο κλάδος αυτός είναι πάρα πολύ δυναμικός και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο το 2017. Ξέρω να τονίσω εδώ ότι η νομοθεσία ε, θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη. Δηλαδή να μην ε, επηρεάζεται από τις εξελίξεις τεχνολογίας, θα πρέπει να ε, καλύπτει με τέτοιο τρόπο ώστε το κόστος και ωφέλεια να είναι ανεξάρτητο από τη τεχνολογία. Στοιχεία νομοθεσίας όπως είναι CCP, CSD και για το Big Data γίνεται πολλή δουλειά αυτό τον καιρό από τις τρεις ρυθμιστικές αρχές για να δούμε ποια είναι τα προϊόντα και πώς μπορούν αυτά να αλλάξουν την προστασία των ε, παιδιτών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που πρέπει να σας διακόπτω, αλλά ε, ο χρόνος είναι δεδομένος. Ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σας αφαιρώ το λόγο. Ο Γκρέκ Βαν Έλσεν. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας παρουσιάσω και εγώ την άποψη του καταναλωτή Η χρηματοπιστωτική τεχνολογία και η ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν ε, τα της ε, οικονομικής του ζωής. Επηρεάζει όμως και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπάρχουν λοιπόν βασικά μηνύματα. Πρώτον, ότι οι αλλαγές ε, είναι ευπρόσδεκτες και χρειαζόμαστε την ε, ψηφιακή αναβάθμιση της προστασίας του καταναλωτή. Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα apps και οι πλατφόρμες δεν λύνουν ε, ε, τα προβλήματα, δεν λύνουν τα πάντα. Η Εφεί λύσει Μπορούν βέβαια να προσφέρουν αλγορίθμου, αλλά παρόλα αυτά οι καταναλωτέ χρειάζονται προστασία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τώρα θα δούμε κάποιε ε, προκλήσεις ε, που αφορούν στον ορισμό στοιχείων της ε, FinTech. Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα η τεχνολογία. Το κόστος της κατανομής μπορεί να προσφέρει να μειωθεί και να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση ε, στους καταναλωτές. Αλλά επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές ερωτήσεις, όπως τι θα γίνει με τους ε, ψηφιακά αναλφάβητους. Αυτοί θα πληρώνουν περισσότερο στο μέλλον για τις ε, ψηφιακές υπηρεσίες ή τι πρόκειται για τις τοξικές επενδύσεις, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχουμε ήδη αναφέρει τους, το crowdfunding, ε, αυτό, αυτή η λέξη είναι της μόδας και μπορεί να είναι και πολύ ενδιαφέρουσα για τους ε, καταναλωτές, ε, όμως αυτό δεν καλύπτεται στην νομοθεσία και υπάρχουν και κάποιες αυθαιρεσίες σχετικά με το crowdfunding. Εξάλλου βλέπουμε και τις ιστοσελίδες όπου γίνονται συγκρίσεις των τιμών και βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ε, πριμ. Αυτό δεν είναι κακό. Από την άλλη όμως όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν και την ποιότητα των προϊόντων. Ε, γιατί υπάρχουν ε, προϊόντα όπου, για τα οποία υπάρχει ιστοσελίδα με τη σύγκριση στοιχείων. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι σημαντικά. Μέχρι τώρα είχαμε τις ε, τράπεζες και τις ασφάλειες ε, που πολύ συχνά ε, πρόσφεραν προϊόντα για να καλύπτουν το κόστος Όλα αυτά είναι ευπρόζεκτα, κυρίως αν μπορούν να ε, εστιαστούν σε συγκεκριμένες ε, υπηρεσίες. Όπως έχουμε δει, παραδείγματο χάρη στον τομέα ε, των διασυνοριακών μοντέλων. Επίσης, τα ρομπότ είναι ενδιαφέροντα για τους καταναλωτές, γιατί μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση σε άλλου είδους συσκευές, και από πλευρά ρυθμιστική έχουμε δύο πλατφόρμες. Η μία δίνει πληροφορίε για τη μύφη, η άλλη όχι. Στον καταναλωτή όμω όλα αυτά μοιάζουν. Άρα δηλαδή αυτό το περιβάλλον είναι μια αρκετά μεγάλη πρόκληση. Και αυτό που αναφέρθηκε και προηγουμένω είναι τα big data ε, τα οποία έχουν, ε, κρύβουν κάποιες, ε, κάποια πλεονεκτήματα, δίνουν περισσότερο προσωποποιημένες, ε, εξατομικευμένες μάλλον πληροφορίες στους καταναλωτές. Αυτό που παίζει ρόλο και θέλω να το προβάλλω είναι ότι βεβαίως και περιλαμβάνονται κινδύνοι μεγαλύτεροι όσον αφορά την ιδιωτική σφαίρα και τον αποκλεισμό. Αν θέλετε, ε, το επίπεδο παιδείας των φίλων μου στο facebook αυτό μπορεί να επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο τη δική μου την ζωή και την σταδιοδρομία την αξιοπιστία το ποσοστό ε, το επιτόκιο δανεισμού και την, τη λήψη δανείου Αυτά, αν θέλετε, είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε και να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον τελευταίο μιλητή μας εξ αποστάσεων, τον Τζέσι McWaters. Thank you so much. Um, it's a great honor to be asked to address this committee. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον, τον Ιανουάριο του 2014 το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξετάζει το πώς τεχνολογίες επηρεάζουν την δομή και διανομή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Κάναμε 300 συνεντεύξεις και πολύ άριθμα εργαστήρια σε ολοκληρωτόν κόσμο για να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Θεωρούμε λοιπόν πως ε, οι καινοτομίε στο FinTech μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες, πιο αποτελεσματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ένα πιο σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όποιος, με οποιαδήποτε καινοτομία όμως υπάρχει κίνδυνος και νέες προκλήσεις. Και βεβαίως θα πρέπει ε, όσοι χαράσουν πολιτική όπως εσείς να προστατεύσουν την δυνατότητα που έχει ο κλάδος. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε τρία συγκεκριμένα τις συγκεκριμένες τομείς που έχουμε παρατηρήσει όσον αφορά την καινοτομία και να προτείνω κάποιες αρχές ορθής διακυβέρνησης με βάση παρατηρήσεις μας. Ο πρώτος τομέας καινοτομίας είναι η μεταμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη. Αυτό βασίζεται κυρίως ε, σε νέες ευέλικτες εταιρείε, οι οποίες έχουν πολύ εστιασμένα επιχειρηματικά μοντέλα και στοχεύουν ακριβώς εκεί πέρα όπου βρίσκεται ή ε, το πρόβλημα πιθανώς ενός πελάτη και τα υφιστάμενα αποθεματικά κέρδους. Έτσι προσφέρουν πολύ πιο εστιασμένες και απλοποιημένες διαδικασίες πληρωμών και θα πρέπει βεβαίως να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και να είναι οι προσφορές τους οι κατάλληλες και δίκαιες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια αρχή η οποία θα είναι μια αρχή ένεργου εμπλοκής και βεβαίως θα πρέπει ταυτόχρονα να βοηθήσουμε την ανάπτυξη θετικών σχέσεων. Η τεχνική αυτή έχει ακολουθεί ήδη με μεγάλη επιτυχία από την CFB στι ΗΠΑ και έχει ακολουθεί μετά και από διάφορε άλλε ρυθμιστικέ αρχέ. Ο δεύτερο κλάδο καινοτομία είναι εντό των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Έτσι δηλαδή αναπτύσσεται μια μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και μειώνεται το κόστος, αλλά αυτό βέβαια δυσκολεύεται από το ότι υπάρχουν κάποια ιστορικά συστήματα στα οποία έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις. Και άρα έχουν κάποιες έχουν εμφανιστεί κάποιες εταιρείε οι οποίες έχουν ακριβώς ως στόχο να υπάρξει μια απλοποίηση των διαδικασιών. Η ορθή διακυβέρνηση βεβαίω θα απαιτήσει σε όσου χαράζουν την πολιτική να δώσουν την δυνατότητα μια ε, καλή συνεργασία. Κάτι το οποίο βλέπουμε παραδείγματο χάρη στην FSA του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ασφαλή χώρο έτσι ώστε μεγάλα και μικρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μπορούν να δοκιμάζουν τα νέα τους και καινοτόμα προϊόντα. Τέλος, ε, όπως ήδη ανέφερε και ο τελευταίος ομιλητής, ε, γνωρίζουμε όλο και περισσότερα τις νέες τεχνολογίες όπως το blockchain που θα μπορούσαν να επανεφεύρουν ολόκληρη την υποδομή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και έτσι υπάρχει δυνατότητα να ξαναχαραχτεί ο χάρτης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, να ανατραπούν οι υποθέσεις οι οποίες αποτελούν τη βάση πολλών επιχειρηματικών μοντέλων και να δώσουν την ε, δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να γίνονται οι εξοφλήσεις ε, σύμφωνα με την ευχέρεια των πελατών. Πιστεύω πως πρόκειται για ευκαιρίες εμφανίζονται μία φορά κάθε γενιά και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο ε, διαφανές δίκαιο και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι και εποπτικές αρχές και εσείς οι πολιτικοί θα πρέπει να αγκαλιάσουν αυτή την ευκαιρία και βεβαίω να έχετε μια ανοιχτή στάση όσον αφορά την αρχιτεκτονική της νέας αυτής υποδομής και βεβαίως να ακούσουμε το τι θα ε, ζητήσουν όσοι δυνατότητες για να μπορέσουν πιο γρήγορα να αντιδράσουν στους νέους κινδύνους που θα προκύψουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη προσοχή. Και τώρα ακολουθεί ο γύρος ερωτήσεων των Ευρωβουλευτών όπως κάναμε και προηγουμένως. Η κόρα πρώτη, <laughs> δεν λέω τίποτα άλλο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές μας και εγώ ε, για τις ενδιαφέρουσες ομιλίες. Μερικά σύντομα ερωτήματα. Ρωτώ το ρυθμιστή, γιατί μιλάτε και εξ ονόματος της ΑΙΟΠΑ και της ε, EBA, της ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Έχουμε τους νέους παίκτες, τους νέους fintech, μικρούς και μεγάλους. Έχουμε και τους μεγάλους που είναι Google και Amazon και τέτοιοι ε, και δραστηριοποιούνται και αυτοί στο συγκεκριμένο κλάδο. Και επειδή η νομοθεσία μας βασίζεται κυρίως σε θεσμούς ε, και ε, διαδότηση των θεσμών αυτών, τι γίνεται με τους ίσους κανόνες παιχνιδιού, αυτό πώς το επηρεάζει. Δηλαδή κοιτάμε περισσότερο τις δραστηριότητες και όχι ποιος τις παρέχει δεν κοιτάμε ας πούμε, τι θεσμός είναι, αν είναι τράπεζα, είναι πληρωμή. Κοιτάμε τη δραστηριότητα αυτή καθ' αυτή και όχι τον πάροχο. Και μια ερώτηση επίσης για τις ρυθμιστικές αρχές και τις εποπτικές αρχές. Τη δικιά σας δουλειά πόσο την επηρεάζει αυτό, γιατί είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από το να είσαι δικηγόρος και να ε, ασχολείσαι με τα νομικά θέματα και άλλο είναι να ψάχνεις αλγορίθμους αν πάει κάτι στραβά. Έχετε το προσωπικό που χρειάζεται για αυτό το σκοπό, έχετε τέτοια στελέχη. Και θέλω να ρωτήσω και τον τελευταίο ομιλητή από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Βλέπετε καμιά διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο ως προς την καινοτομία, ε, το οικοσύστημα αυτό εμείς είμαστε πρωτοπόροι, υπολοιπόμεθα, έχουμε μείνει πίσω, πρέπει να επιταχύνουμε, είμαστε εντάξει, μπορεί να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστές η κυρία Μπερές. Α, συγγνώμη, όχι, όχι. Έχουμε μεγαλύτερη ομάδα. <laughs> Ο Μπράιαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα συναρπαστικά τα όσα ακούσαμε και από τους τρεις. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Βανέλσεν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που έθεσε το ερώτημα. Για πάρα πολύ κόσμο που μπορεί να μείνει στο περιθώριο αυτής της επανάστασης. Κάποιος είπε προηγουμένως ότι 9 εκατομμύρια ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν καμία πρόσβαση στις νέες αλλαγές ε, στο τραπεζικό σύστημα ε, πρόσφατα. Και μετά είπε ότι ένα από τα αρνητικά θα μπορούσε να είναι αυτό, ότι ε, μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες θα χρεωθεί περισσότερο τις παραδοσιακές. Και ρωτώ, πού είναι η ευθύνη εδώ του κλάδου ή που θα έπρεπε να βρίσκεται όταν πρόκειται Γι' αυτό. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι δεν θα μείνουν στο περιθώριο πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω αυτών των ριζικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Ποιος είναι αρμόδιος, το κράτος, η Ευρώπη, ο ίδιος ο κλάδος δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει προσπαθώντας να εξασφαλίσει να μην αφαιθούν στην άκρη κάποιοι άνθρωποι και να έχουν και αυτοί τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Ακόμα και αν είναι ψηφιακά αναλφάβητη και δανείζομαι τη δική σας έκφραση. Ευχαριστώ. Τώρα όμως η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις έχω. Πρώτον, προφανώς η αφετηρία για όλη αυτή τη συζήτηση είναι η ιστορία των πληρωμών. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλές άλλες εξελίξεις οι οποίες παράλληλα ε, μπορούν να βασιστούν σε αυτή τη στρατηγική καινοτομίας ε, με τις κρυπτογραφημένες τεχνολογίες. Αυτό που με ενδιαφέρει μένα είναι η διαφοροποίηση και η ποικιλία των υπηρεσιών. Και μετά έχουμε αυτή την τεχνολογική καινοτομία που προφανώς πρέπει να την αφήσουμε να αναπτυχθεί και από την άλλη εμείς έχουμε κάποιες εργασίες για την οδηγία για την καταπολέμηση της ε, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, anti-money laundering, ε, το ξέπλυμα κοινώς εμείς οι νομοθέτες ε, θα πρέπει ίσως από αυτό το στάδιο ήδη να παρέμβουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε σε λάθος κατεύθυνση ή στην αντίθετη από την επιθυμητή, ε, από αυτή που αποσκοπεί ο νομοθέτης, εμείς δηλαδή. Και ένα τελευταίο από τον εκπρόσωπο της ε, BUC εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία σας. Έχουμε και πολλές αναφορές που έρχονται εδώ στην Επιτροπή Αναφορών και ε, απορρέουν από πολίτες που έπεσαν θύματα απάτης. Ε, γιατί απάντησαν ε, σε διάφορα κλικ που τους έταζαν λαγούς με πετραχίλια και τους πήραν τα λεφτά από τους λογαριασμούς τους. Εσείς τι κάνετε ως BUC δύο-τρία συγκεκριμένα πράγματα, τέσσερα ξέρω εγώ, όχι για να τα επιβάλλουμε, αλλά για να προσπαθήσουμε να τα ε, ε, εντάξουμε στην νομοθεσία μας. Τι θα κάνουμε, αυτό αφορά τις εποπτικές αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές. Τι λέει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. ECR, ο κύριος Φόξ. Uh, thank you, President. Can I thank the speakers for... Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ομιλητές ε, για τις ομιλίες τους. Θα γνωρίζετε ότι στο Ηνωμένο Βασιλείο ο ρυθμιστής ε, έχει βάλει ένα ανάχωμα. Διερωτώ με λοιπόν ε, κατά πόσο το έχετε αυτό εξετάσει. Γιατί εάν υπάρχει ή αν υπήρχε εδώ στην Ευρώπη, πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο το έβαλε αυτό μόνο του, το ανάχωμα, ας πούμε, τη Σιγκαπούρη και τα πράγματα πάνε καλά. Και ρωτώ, ε, θα μπορούσαν να συνενωθούν τα κέντρα της FinTech ή θα υπήρχε μια τελείως άλλο διαφορετική προσέγγιση. Κάτι άλλο. Τι είναι εκείνο που εμποδίζει την Ευρώπη να ε, αυξηθεί ακόμα, να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να ανταγωνιστεί τελικά το Silicon Valley. Περίπου ε, σε αυτό το κανάλι, σε αυτή τη διεύλο θέλω να συνεχίσω και εγώ, δηλαδή πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή και τι είδου ε, μέτρα μπορούμε να προτείνουμε έτσι ώστε να τα εφαρμόσουμε και στα 28 κράτη-μέλη και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ε, γρήγορος και αποτελεσματικός. Προηγουμένως είπα ότι φοβάμαι ότι με μεγαλύτερη ευελιξία στα προϊόντα fintech θα δημιουργηθούν νέα προβλήματα τα οποία δεν είχαμε στα κλασικά τραπεζικά προϊόντα με το χαμηλότερο κόστος συναλλαγής και με τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Παρακαλώ, οι παρακαθήμενοι σας, ευχαριστώ και εγώ. Εγώ μία σύντομη ερώτηση δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός ορισμός ε, για το FinTech. Εσείς ε, έχετε έναν ορισμό για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτά τα FinTech. Θέλετε εσείς ε, συγκεκριμένο ορισμό. Και να το πω και αλλιώς, δεν είναι επικίνδυνο να θέλουμε να μαθητήσουμε κάτι που καταρχήν δεν έχουμε ορίσει με ακρίβεια. Πολλές ερωτήσεις από ό,τι βλέπετε, άρα και εμείς περιμένουμε πολλές απαντήσεις. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, και στις δύο ερωτήσεις της ε, κόρας ε, και σε μία ερώτηση κυρίας Περές. Πολύ σωστά λέτε ότι μας ενδιαφέρει η προστασία του καταναλωτή Εκεί θέλησαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας και τελικά ε, καταλήξαμε σε άλλους κανόνες που έχουν σχέση και με τις ασφάλειες ε, ε, και με τον επιμερισμό των ασφαλιών. Εμείς προσπαθήσαμε να τα ξεδιαλύνουμε όλα αυτά και σε ευρωπαϊκό και δυνατόν και σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της ε, AMLD θα συμφθεί μετά από λίγους μήνες μια κοινή γνώμη για το πώς αξιολογούνται οι κίνδυνοι στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Και θα δείτε ότι αυτή η γνωμοδότηση δεν βασίζεται τόσο στην ε, κοινωτική νομοθεσία, αλλά στο πώς ε, μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μπορεί να προκύψει μετά από κάποια χρόνια. Το άλλο θέμα που θέλω να δείξω είναι πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε ανάμεσα στους μεγάλους και τους μικρούς παίκτες. Εδώ τίθεται και το θέμα της ε, αναλογικότητας ε, και σε σχέση με τους συνομοθέτες, ε, την εποπτεία. Θα έλεγα ότι πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς προκαταλήψεις και θα έλεγα ότι οι ρυθμιστές πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο στην εποπτεία της FinTech χωρίς προκαταλήψεις. Όσον αφορά στην ερώτηση σχετικά με το ε, ευρωπαϊκό ανάχωμα, Εμείς όταν μιλήσαμε για το crowdfunding είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν βασικοί κανόνες για το crowdfunding γιατί ήταν ε, μία από τις πρώτες συγχωνεύσεις στην Ευρώπη. Αυτό δεν έγινε, αλλά για να υπάρχει έτσι ένα τέτοιο ε, ανάχωμα, νομίζω ότι Αυτή είναι μια πολύ φιλόδοξη προσέγγιση από ευρωπαϊκή σκοπιά για να θελήσει κανείς να συστήσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι όσον αφορά τους καταναλωτές, ε, τους μικρούς επενδυτές, ε, αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα πολλών προϊόντων και κάπου τα έχουν χαμένα. Έχουν χάσει, γιατί τα έχουν χάσει, δεν υπάρχουν και καλές προτάσεις για αυτού του είδους τους καταναλωτές. Εμείς ε, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό των ε, καταναλωτών δίδοντάς τους περισσότερες πληροφορίες, ε, καταρτίζοντας κανόνες οι οποίοι διαφέρουν αλλιώς τις ασφάλειες, αλλιώς τις τράπεζες και αλλιώς αυτούς που χειρίζονται κεφάλαια. Είναι ένα πολύ περίπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αν έχει κανείς κατά νου διάφορες χρηματοπιστωτικές ανάγκες, αν έχει κατά νου τυποποιημένα προϊόντα για τους ε, καταναλωτές, αυτό μπορεί να δημιουργήσει την άποψη ότι ως ε, καταναλωτής ε, είτε θα πάει κανείς για τις στάντα λύσεις, είτε θα βγει έξω από την προστατευμένη περιοχή. Άρα δηλαδή σε γενικές γραμμές αυτό παρατηρεί κανείς. Και το δεύτερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε καλύτερη εποπτεία και με τους ισχύοντες ε, κανόνες, ε, παραδείγματος χάρη σχετικά με τα MIFID, ε, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι θα ενημερώνονται σωστά. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να ληφθούν υπόψη. Φίντεκ μπορεί να βοηθήσει μπορεί να βοηθήσει ε, στο να υπάρχουν απλά προϊόντα για τους ε, καταναλωτές. Και αυτό μπορεί να το επιτύχει η ψηφιοποίηση. Uh, um, Προσπαθήσω να απαντήσω γρήγορα. Είναι πάρα πολύ κακός ο ήχος και δεν μπορούμε δυστυχώς να τα μεταφράσουμε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 Τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσει. Παρακαλώ, κόρα. Σύντομα. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση, συναρπαστική θα έλεγα και επίσης μας δώσατε ε, τροφή για σκέψη. Και ε, προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους σκιώδεις ηγητές για την έκθεσή μου. Γιατί αν έχουμε προϊόντα που είναι ταχύτερα, φθηνότερα, καλύτερα, γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε στην Ευρώπη και γιατί να μην είμαστε κι εμείς ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστούμε και πάλι που μας ήρθατε και θα παραμείνουμε σε επαφή με όλους σας στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ όλους σας. Συνεχίζουμε στην ημερήσια διάταξή μας κανονικά.

Excuse me, if you don't mind, we'll try to continue with the, with the committee. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Παρακαλώ, ηρεμήστε. Okay, Continuamos. Συνεχίζουμε λοιπόν, σας παρακαλώ. Ησυχία. You go to speak. Yes. Please go out. Παρακαλώ, ιδιωτικέ συνομιλίε εκτό τη αιθούση. Τα λεγόμενα πηγαδάκια, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε. Δεν τελείωσε η Επιτροπή. Thank you. Continuamos ahora con el punto. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στην ημερήσια διάταξη θέσπιση είναι το σημείο 12. Έλεγα λοιπόν θέσπιση ενωσιακού προγράμματο για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση τη συμμετοχή των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακή πολιτική στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσω αμέσω το λόγο στο Φιλίπ Λάμπερτ, στον εισηγητή μα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ βεβαίως τη μεγάλη προσέλευση ε, για τη χρηματοδότηση του Finance Watch. Χαίρομαι που σας ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με βοηθάτε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Mm. είμαι και επικεφαλής ομάδας. Λοιπόν, θα μιλήσω στα αγγλικά. Λοιπόν, πρόκειται για μικρή αλλά σημαντική πρωτοβουλία. Πρόκειται για χρηματοδότηση οργανώσεων όπως το Finance Watch και Better Finance, αποτέλεσμα διακομματικής πρωτοβουλίας στην προηγούμενη θητεία και θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συνένεση. Αργήσαμε λίγο, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. με την έννοια ότι υποστηρίζουμε σε γενικές γραμμές ε, την πρόταση της ε, Κομισιόν για να έχουμε μια μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και να μπορούν οι οργανώσεις αυτές να έχουν κάποιο βαθμό σταθερότητας. Δεύτερον, να καθορίσουμε τις δύο αυτές οργανώσεις που είπα Better Finance και Finance Watch που ήταν αυτές που έκαναν πρώτες αίτηση δεν είναι δηλαδή ότι μας αρέσουν καλύτερα Αυτές ανταποκρίθηκαν καλύτερα στην πρόκληση όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία και τέλος βεβαίως το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος καθώς δεν αφορά μόνο την έρευνα και την ενημέρωση αλλά και την στήριξη των θέσεών μας. Δεύτερον, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο περιορίσαμε τις τροπολογία είναι για λόγους ταχύτητας για να τελειώνουμε το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε οι οργανώσεις να έχουν το 2017 μια σωστή βάση. Μετά οι τροπολογίες είναι περιορισμένες, σε δύο αφορούν το πεδίο εφαρμογή για να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητε πολιτικής αλλά και συμβουλευτικής υπηρεσίας να καλύπτονται αλλά βεβαίως και όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού για τους σχετικούς κανονισμούς. Έχουμε επίσης μια τροπολογία για τους στόχους του προγράμματος που αναφέρονται στους στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το πολυμερές επίπεδο, G20, ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας, καθώς παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό προδιαγραφών που αργότερα γίνονται ευρωπαϊκό δίκαιο και θα πρέπει να παρεμβαίνουν νωρί στην διαδικασία όταν δηλαδή συζητούνται αυτές οι προτάσεις ε, παρουσία των ε, ξεματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τώρα αυτή την εβδομάδα στην Χιλή. Μετά Έχουμε μια τροπολογία στο άρθρο 3 το οποίο αφορά τις απαιτήσει για τους δικαιούχους για να μην υπάρχουν λοιπόν συγχύσεις μεταξύ του προγράμματος της Κομισιόν και των δραστηριοτήτων προτείναμε η παράγραφος 2 του άρθρου 7 να πάει στο άρθρο 3 το οποίο αφορά τις απαιτήσει από τους δικαιούχους συγκεκριμένα σύμφωνα με το εκτιμώντας 14 της πρότασης της Κομισιόν προτείναμε σε μια νέα παράγραφο οι δικαιούχοι να υποβάλουν σε αιτήσια βάση μια περιγραφή των δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος. Και έτσι θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς οι δραστηριότητες, οι στόχοι, το κόστος και οι σχετικοί δείκτες αξιολόγησης. Γιατί κάναμε κατεύθυνση. Κοιτάξτε, η τροπολογία αυτή είναι κάτι παρόμοιο με αυτό το οποίο έκανε η κυρία Φόρντ στην ΙΜΚΟ και έτσι βεβαίως θα έλεγα ότι τίνουμε και μια χείρα φιλία στην ΙΜΚΟ αλλά το να μετακινηθεί αυτό το άρθρο από το 7 στο 3 θα διαχωριζόταν το πρόγραμμα της Ένωσης από το πρόγραμμα των οργανώσεων αυτών. Να μην έχουμε δηλαδή το πρόβλημα που τονίσαμε πριν ότι εφόσον τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν παρέχουν το 100% της χρηματοδότησης σωστό είναι να μην καθορίζουν 100% το πρόγραμμά τους. Δηλαδή, να μην καθορίζει ολόκληρο το πρόγραμμά τους η Κομισιόν με μερική μόνο χρηματοδότηση. Όποιος ε, πληρώνει δηλαδή αποφασίζει. Αυτό ήθελα να πω. Αυτά να ακούσουμε και τους σκιοσυγητές για να τελειώνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάμπερτς. Οι διάφορε σκιώδεις λοιπόν ακολουθούν. Από το Λαϊκό Κόμμα η κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας. Ε, πολύ ισόρροπη προσέγγιση στην έκθεσή του, ε, πάρα πολύ καλή πάρα πολύ εύστοχη και όχι μόνο επί της αρχής αλλά και τεχνικά είναι από τις πιο δύσκολες εκθέσεις που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπως είπε και ο ίδιος το 2010 άρχισε αυτή η προσπάθεια ε, διακομματικά συμμετείχαν οι συντονιστές των μεγάλων πολιτικών ομάδων έτσι ώστε να αρχίσει αυτή η προσπάθεια ε, να καταλάβουμε τι γίνεται ε, σε αυτό το τομέα της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητα. Οπότε είναι επόμενο και μοιραίο ότι συνεχίσαμε την προσπάθεια αυτή. Είναι αποδεκτές οι τροπολογίες. Η τρία είναι κυρίως ε, τεχνική, αλλά για να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις, πώς να το πω, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ νομίζω πρέπει να αλλάξει αυτό και να χρηματοδοτείται από την αγορά. Για τους καταναλωτές είναι πάρα πολύ σημαντική προστασία. Γενικά συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστές, ο κύριος Λούτβιξον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω την πρόταση της Επιτροπής ε, για κανονισμό και ε, θεωρώ ότι πρέπει να υποστηριχτούν όλες αυτές οι δραστηριότητες. Η πρωτοβουλία για τα πιλωτικά προγράμματα που ξεκίνησε η Κομισιόν ε, το 2011 επέτρεψε να υπάρξει βελτίωση των οικονομικών ε, γνώσεων, των τεχνοοικονομικών γνώσεων και να ε, μπορέσουν οι καταναλωτές ε, να εμπλακούν στα προγράμματα αυτά. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και θεωρώ ότι πρέπει να διευκολυνθεί η θέση των Ευρωπαίων πολιτών να τοποθετούνται επί της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας γιατί αυτό που λείπει είναι η επαρκή πόρη έτσι ώστε να εμπλέκεται κανείς, να μπορεί να συμμετέχει σε πολύ ε, τεχνικές συζητήσεις που έχουν σχέση με την νομοθεσία, στο, κυρίως στο θέμα των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, πολλές δυνατότητες. Ε, πολλοί θα πρέπει να απελευθερωθούν από, τον, από τις επιρροές και να είναι ανεξάρτητοι και είναι πολύ σημαντικό αυτή η φορείς, ε, συγγνώμη, θα πρέπει να δουλέψουν σκληρότερα έτσι ώστε οι διατάξεις να είναι πολύ πιο εύκολες για, τους, για την κοινή γνώμη οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να συμμετέχουν στην καθημερινή εργασία των νομοθετών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε νέες μεθόδους ε, που να λειτουργούν σωστά και τελικά, αν αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα πρόκειται να γίνει πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της Επιτροπής. Η Beta Finance και η Finance Watch θα πρέπει να συμμετέχουν καλύτερα στην ε, ανεξαρτησία από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εμπιστοσύνη του κοινού εξαρτάται από τους εξωτερικούς ε, παράγοντες. Αυτοί λοιπόν οι οργανισμοί πρέπει να αναζητήσουν την πλήρη ανεξαρτησία από τους ε, θεσμούς. Ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, σχετικά με την εμπλοκή διαφόρων συμφερόντων. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για τους οργανισμούς αυτούς να χρηματοδοτούνται από οποιονδήποτε άλλο πέρα από τον χρηματοψηφιακό κλάδο. Ε, θα, συνεχίσουμε το πρόγραμμα από το 14 έως το 20 και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό για το δημόσιο συμφέρον. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι εγώ στηρίζω πλήρως τον εισηγητή σε όλα αυτά που είπε και ελπίζω ότι θα καταστεί δυνατό να βρούμε μια καλή λύση από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. <laughs> Ο κύριος από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν φύγει από την αίθουσα θα ήθελα να συγχαρώ επ' ευκαιρία τον νέο μας αντιπρόεδρο, ο οποίος και μιλάει και ισπανικά και παρόλο που είναι από τα Κανάρια νησιά και ξανθός, είναι πολύ καλός μου φίλος. Ε, και θέλω να πω τα βασικά. Η ομάδα μου θα υποστηρίξει τη συνέχεια ε, στη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέπεια για τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων. Έχουμε επίγνωση ότι ε, ούτως πράττοντες υποστηρίζουμε την καλύτερη υπηρεσία προς τους καταναλωτές και ταυτόχρονα και την ανεξαρτησία και μάλιστα ανεξαρτησία κατά του λόμπι που είναι ε, απολύτως απαραίτητη σε ένα πλουραλιστικό κόσμο. Τον των τέσσερα είναι τα θέματα για μας που είναι σημαντικά. Πρώτον, τα χρήματα θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν αφιβάλλω καθόλου για την ακαιρεότητά τους, γιατί έχει γίνει τώρα μια μεγάλη φασαρία, ε, μεγάλος άλλος στην Όλαφ και τα λοιπά. Ε, καμία σχέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει δικαίωμα, πιστεύω, να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει ε, στο ετήσιο πρόγραμμα ή σε ένα τμήμα του και ακόμα και να ελέγχει τα προγράμματα. Καλά, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα χρηματοδοτεί όλα. Είναι θεματοφύλακα των συνθήκων. Δεν μπορεί να χρηματοδοτεί ένα κείμενο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φερρυπίν. Εδώ όμω υπάρχει ένα θέμα και η πρόταση του κύριου Λαμπέρτς πηγαίνει στην καλή σωστή κατεύθυνση. Εμεί μπορεί να κάνουμε καμιά τροπολογία για να το διευκρινίσουμε. Ένα δεύτερο θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι έχουμε μπει σε νέα φάση τώρα της χρήσης ε, των ε, δύο εταιριών ή οργανισμών. Έχει φτάσει η ώρα όπου, πώς να το πω τώρα, Μπράβο, πολύ ωραίο το τριετές πρόγραμμα γιατί έτσι να υπάρχει και μεγαλύτερη ανεξαρτησία και πολύ καλύτερα θα γίνεται η δουλειά με μεγαλύτερη σοβαρότητα και δεν θα χανόμαστε ε, τα βραχυπρόθεσμα και ε, επίσης δεν θα πλατιάζουμε κιόλα. θα πρέπει να είναι στοχευμένη η δουλειά ε, και εδώ θα κάνουμε μια πρόταση, θα διαβάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά τι λέει η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για την προστασία των καταναλωτών και αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι δύο αυτοί οι οργανισμοί δεν κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ο ένας βρίσκεται πολύ πιο κοντά στους καταναλωτές και στην κοινωνία των πολιτών και η άλλη είναι ερευνητικό κέντρο με την αυστηρή έννοια που ελέγχει και αξιολογεί εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. Και οι δύο οργανισμοί είναι σεβαστοί, αλλά θα κάνουν τροπολογίες ζητώντας να κάνουν μια προσπάθεια και να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάδοση. Γιατί έρχεται μια στιγμή που μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει αυτά και να τα αξιοποιήσει, ας πούμε με τα διάφορα γραφεία που έχει σε διάφορα κράτη-μέλη. Ε, τα κέντρα, πώς τα λένε αυτά, ενημέρωσης για να φτάσει σε όλες τις γωνιές η πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μέχρι τώρα η δουλειά που ήταν, ε, το ήταν πολύ βραχυπρόθεσμη και πάρα πολύ τοπικού χαρακτήρα και δεν βοηθούσε καθόλου ορισμένε χώρες. Θα μπορούσαμε ε, να βοηθήσουμε και με τροπολογίες. Γενικά συμφωνούμε λοιπόν, αυτά ήταν τα θέματα που ήθελα να αναφέρω. Βέβαια θαυμάζω πάρα πολύ τον κύριο Λάμπερτς και τον Τιμό και από την ΙΜΚΟ θα δούμε λοιπόν τι θα πει εκεί η δική τους ε, συντάκτρια γνωμοδότησης και θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ, ο Ματ Κάρθη. Thank you, Chairman, and thanks to the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και, και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ε, γενικά συμφωνούμε με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την έκθεση και με όλες τις τροπολογίες του εισηγητή. Υπάρχουν κάποια σημεία που θα θέλαμε ε, να δούμε στην τελευταία τελική έκθεση. Χρειαζόμαστε καλύτερη χρηματοδότηση ε, και όχι μόνο παροχή συμβουλών ε, είναι περίπλοκα τα θέματα και χρειάζονται βοήθεια καταναλωτές. Ε, είναι πολύ τα προβλήματα γνωρίζουν οι περισσότεροι ε, ευρωβουλευτές και έχουν επωφεληθεί προσωπικά από την παροχή συμβούλων. Επίσης, θα πρέπει οι οργανώσεις να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά, δηλαδή να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών στο κοινό σε πλήρη ανεξαρτησία να δρούν ως προς τη χρηματοδότηση από τα θεσμικά όργανα. Δηλαδή, αυτά που καλύπτουν και τα αποτελέσματα των ερευνών ε, πάντα ε, δεν θα ικανοποιούν τους πάντες, μα αυτό είναι ορισμός της ανεξαρτησίας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αλλιώς έχει εξυπηρετήσει ιδιωτελή συμφέροντα και είσαι κατευθυνόμενος. Ε, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απολύτως ανεξάρτητα να παράγουν τα αιτήσια έγγραφά τους. Αυτά θέλαμε να δούμε στην τελική έκθεση και προσβλέπουμε συνεργασία με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους και όλους εισηγητές. Ευχαριστώ. Thank you, uh, von Ευχαριστώ, η Beatrix von Storch. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισηγητά. Μεγάλη ομοθυμία βλέπω εδώ αλλά και την τελευταία φορά εγώ είχα ε, εκφράσει τις αμφιβολίες μου και δεν έχω αλλάξει πάρα πολύ άποψη. Δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί θα πρέπει να χρηματοδοτούμε ε, το Finance Watch και το Better Finance που είναι λόμπι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχει νόημα ως κοινοβούλιο να πληρώνουμε οργανώσεις που έρχονται μετά να μας συμβουλεύουν για την νομοθεσία μας, για τα συμφέροντα των καταναλωτών. Έχουμε κάθε δυνατότητα στο Κοινοβούλιο έχουμε δυνατότητες ε, να απευθυνόμαστε σε think tanks, έχουμε χρήματα από το Κοινοβούλιο, έχουμε τεχνογνωσία στις πολιτικές ομάδες και μια σειρά άλλες δυνατότητες. Έχουμε δικούς μας υπαλλήλους, συνεργάτες Έχουμε Ινστιτούτα δημόσια ή μη και δεν συμμαζεύεται που μπορούμε να ανατρέχουμε. Για ποιο λόγο λοιπόν θα πρέπει ο καταναλωτής, όχι μάλλον ο φορολογούμενος, να πληρώνει 6 εκατομμύρια χρήματα σε οργανώσεις λόμπι. 6 εκατομμύρια ευρώ είναι από το 2017 μέχρι το 2020. Για ποιο λόγο να τα επιβαρυνθεί αυτά ο, ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Γι' αυτό έκανα τροπολογία για να καταργηθεί αυτή η χρηματοδότηση και θα χαιρόμουν να με υποστηρίζετε. Ευχαριστώ. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί μας. Ο κύριος Σάλλας, παρακαλώ. Σάλλας. Chairman, colleagues, good afternoon. Uh, I will try to, to, to be uh, brief. Uh, first of all, I would like to thank... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαιρετικό του έργο στην πρόταση αυτή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, ευχαριστώ και τους υπόλοιπους και για τα καλά τους σχόλια. Στόχος της πρότασης ε, ήταν αυτός που συνόψισε ο κύριος Λαμπέρτς και ο κύριος Λούντβιξον, οπότε δεν πρόκειται εγώ να επεκταθώ σε αυτό. Ε, ένα-δυο σχόλια ή προτάσεις να σχολιάσω κι εγώ. Δεν έχω δει ακόμα τα σχέδια τροπολογιών για την περιορισμένη διάρκεια του προγράμματος εργασίας και ε, το άρθρο 7 και 3 του εισηγητού εξ όσων καταλαβαίνω. Συμφωνούμε με τους στόχους σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να χρειαστεί να ελέγξουμε κατά πόσο αυτές οι αλλαγές συνάδουν με ε, τους χρηματοπιστωτικούς ε, κανόνες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε ό,τι αφορά ε, τα σχόλια του κυρίου Καλφέ σας επιβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί αυτά τα προγράμματα, έχει αναλάβει την εκτέλεσή τους και ε, θα προσέξει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο δαπανά αυτά τα κονδύλια. Όπως είχα την ευκαιρία να εξηγήσω και στο παρελθόν, δεν θα έχουμε λόγο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια του προγραμματός της, αλλά μια γενική έποψη και πριν προχωρήσουμε στην τελική πληρωμή να ελέγξουμε αν έχουν ανταποκριθεί στο στόχο τους. Όλα αυτά στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής δράσης και του πιλωτικού προγράμματος ε, και είμαι βέβαιος ότι και με τη νέα δομή θα λειτουργήσει καλά. Γενικά σας ευχαριστούμε. Η Επιτροπή σας εργάστηκε πολύ γρήγορα και ελπίζουμε και το Κοινοβούλιο να ε, προχωρήσει μετά την έγκριση και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Γιατί όπως είπε ο κ. Λάμπερτς, καλό θα ήταν στις αρχές του 2017 να είναι δεδομένη η νέα χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, τώρα θα κάνει ο κύριος Λάμπερ το τελευταίο σχόλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους ε, που θέλουν να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι θα τη στηρίξουν οι περισσότερες πολιτικές ομάδες. Καλό αυτό. Και ακούσαμε όλοι ότι η κυρία Βαν Στόρχ ε, θεωρεί ότι όλα αυτά είναι περίτα. Αλλά τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, είσαστε μειοψηφία και φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ε, κάποια συμβαστική πρόταση ανάμεσα στο να συνεχίσουμε και να σταματήσουμε. Ε, θα συνεχίσουμε και να σας πω ένα πράγμα, ότι Τη δική μου την ορολογία, τα λόμπι, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι υπερασπίζονται συγκεκριμένα συμφέροντα. Και αυτό δεν είναι κακό, ε, αλλά πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν συγχαίω τα λόμπι με οργανισμούς οι οποίοι ε, είναι όπως το Finance Watch ε, που προσπαθούν να υπερασπιστούν το τι είναι καλό για την κοινωνία. Αυτοί δεν έχουν κανένα όφελο. Ε, εγώ ποτέ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη λόμπι για αυτού του οργανισμού. Μπορεί κανεί να επιτιμεί αυτοί οι οργανισμοί να χρηματοδοτούνται από ενθουσιασμένου ε, πολίτε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα μέχρι εκεί. Εγώ πιστεύω ότι κάποια μέρα έτσι ήταν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, ω ε, ευρωπαϊκοί θεσμοί λειτουργούμε λιγάκι, λειτουργούμε λιγάκι ως άγγελοι των επιχειρήσεων, βοηθάμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτά. Και είμαι σίγουρος ότι ε, θα καταλήξουμε ε, σε κάποιους ε, συμβιβασμούς για τις διαφορές μας με την Κομισιόν. Θα δούμε τι θα γίνει με τους κανόνες. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να σεβόμαστε τους κανόνες. Ευχαριστώ. 8 Δεκεμβρίου προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι. Στις 12 Ιανουαρίου θα συζητηθούν, ε, θα ψηφιστούν στις 25 του Γενάρη εδώ στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Σας ευχαριστώ. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα consideration. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική ανταγωνισμού. Εισηγητή ο, ο κύριος Τιμπορζάνη. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα δεν είναι θέμα ευγένεια, αλλά ειλικρίνεια. Ναι, ε, τα αλήθεια λέει, το εννοώ αυτό. Να ευχαριστήσω και όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές όλους όσους συμμετείχαν στην σύνταξη της γνωμοδότησης και συνεργαστήκαμε αρκετά καλά τις τελευταίες μέρες επικοδομητικά θα έλεγα μέχρι στιγμής είχαμε λοιπόν εδώ πέρα δύο πολύ αποτελεσματικές συναντήσεις των σκιωδών και προσπαθήσαμε να περιλάβουμε τις απόψεις των διαφόρων ομάδων και βεβαίως τις απόψεις που περιέχονται στην γνωμοδότηση που είχαν εγκρίνει οι άλλες επιτροπές και η Επιτροπή Γεωργίας. Οπότε Είμαι ευγνώμων ε, για το επικοδομητικό αυτό έργο και βέβαια για το ότι οι συνάδελφοι ήταν στην διάθεσή μας. Ε, αν και ομολογώ δεν μπόρεσα να τους συναντήσω όλους. Αλλά νομίζω συνάντησα τους περισσότερους που είναι αρμόδιοι για αυτό το θέμα. Μια άλλη παρατήρηση που ίσως διαφέρει κάπως από άλλες περιπτώσεις όπου η εισηγητής ε, θέλει να υπάρξει κάποια μάχη γύρω από διάφορες εξαιρετικές ιδέες ε, μένα δεν με ενδιαφέρε να κερδίσω κάτι τέτοιο αλλά προσπάθησα να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ε, το Κοινοβούλιο βλέπει την κατάσταση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Λοιπόν, το σχέδιο έκθεσης βασίζεται σε έξι κεφάλαια. Πρώτο και σημαντικότερο, από τη σκοπιά του ανταγωνισμού έχουμε την ε, ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Το δεύτερο, το θέμα της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς. Τρίτον, ένα πολύ επίκαιρο θέμα επίσης, το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Τέταρτον, παραδοσιακές διαδικασίες, αντιτράστ, καρτέλ κτλ. και συγχωνεύσεις. Πέμπτον, τομέακες κλαδικές πτυχές όπως ενέργεια, γεωργία κτλ. Εκτών, ο τομέας των εθνικών αρχών ανταγωνισμού που συχνά απασχολεί και την Κομισιόν και συνολικά προσπάθησα και προσπαθήσαμε με τους σκιώδεις συγητές να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος το πώς θα ενισχύσουμε τον δημοκρατικό χαρακτήρα των πολιτικών συνοχής. Οπότε, θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία τώρα. Χάρηκα ιδιαίτερα που έλαβα τόσες πολλές τροπολογίες από τους συναδέλφους. Συνολικά επέβαλαν 439 τροπολογίες Πάντα το πρώτο σχέδιο βεβαίως είναι κάτι το σύντομο γιατί έχει τα όρια του όσον αφορά το μήκος αλλά νομίζω πως οι τροπολογίες αυτές μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να δούμε το περιεχόμενο του φακέλου. Τώρα, συνολικά έχουμε 27 συμβιβαστικές ε, προτάσεις αλλά πρέπει να ξέρετε ότι κάποιες από αυτές είναι ακόμα υπό συζήτηση με τους σκιώδεις συζητητές οπότε νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα λάβουν τον κατάλογο αμέσως μετά από τη συνεδρία αυτή και ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα στα οποία θα έχουμε μια καλή ισορροπία ικανοποιητική για όλους. Βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε τις πολιτικές προτεραιότητες των διαφόρων ομάδων και μπορώ να σας πω πως και εγώ ως εισηγητής έχω μεγάλη ευαισθησία ε, απέναντι στις προτάσεις των συναδέλφων. Υπήρχε ένα αίτημα που είχα αντιληφθεί από κάποιες πολιτικές ομάδες για να έχουμε μια επανεξέταση της φορολογίας. Να σας δώσω δύο ακόμα παραδείγματα που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί μου στις τροπολογίες. Έχω λάβει πάνω από 50 τροπολογίες που αφορούν άμεσα το θέμα της φορολογίας. Έχουμε γύρω στις 40 τροπολογίες για την γεωργία και λίγο περισσότερες για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Οπότε... Δεν πρέπει να παραπλανηθούμε εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι ζητήματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό. Και ακολουθήσαμε την σωστή νομίζω πορεία. Υπάρχουν βεβαίως κάποια επίμαχα ζητήματα. Ξέρετε νομίζω πως ε, δεν είναι τίποτα φοβερό να πω εδώ στο Κοινοβούλιο ότι ο βασικός μας στόχος είναι μια, ολοένα στενότερη ένωση. Οπότε όταν μιλάμε για διάφορες ενώσεις ε, και η Δημοσιονομική Ένωση δεν πρέπει να είναι κάτι περίεργο. Αν και αντιλαμβάνομαι τις επιφυλάξεις ε, κάποιων ε, συνάδελφων. Αυτό η τωρινή μορφή της έκθεσης δεν ακλά καλύτερα τις απόψεις του Κοινοβουλίου και όχι μόνο μερικών πολιτικών ομάδων. Κάποιοι από μας ή εσάς είχαν κάποιες ε, επιφυλάξεις για το κοινωνικό ντάμπινγκ, αλλά νομίζω ότι το θέμα αυτό πρέπει ακριβώ να το δούμε όπως ακριβώς το είδε το κοινοβούλιο οπότε εγώ δεν βλέπω λόγο να γίνει κάπως διαφορετικά και Ίσως το τρίτο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω δεν κάπως έτσι δύσκολα ζητήματα αφορά το γνωστό, τη γνωστή αυτή πρακτική που κατονομάζουμε τους φταίχτες. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε εδώ μια ισορροπία γιατί ε, υπήρχαν πολλά αιτήματα που έλεγαν ότι χωρίς να κατονομάσουμε υπήρχαν περιπτώσεις αλλά χωρίς να κατονομάσουμε κανέναν θα ήταν πολύ γενικόλογα τα πράγματα αλλά ταυτόχρονα αναφέρουμε ελάχιστες συγκεκριμένες ε, εταιρείες γιατί είπαμε ότι ε, δεν θα ήθελα να γίνει, να γίνει χρήσος οδηγός η έκθεση τέλος κάποιες πολιτικές ομάδες είχαν και κάποιες επιφυλάξεις για την αναφορά συγκεκριμένων καταστάσεων απομακρυσμένων περιοχών. Ε, μετά από συζητήσεις νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τους καλύτερους συμβιβασμούς ε, για όλες τις ομάδες και να συζητήσουμε και αυτά τα πράγματα και αύριο. Έχουμε λοιπόν διαφορετικά σημεία στα οποία συμφώνησαν οι ομάδες σε κινήτες. Δηλαδή φορολογία, εκθέσεις αναχώρα, ενιαία αγορά, ανταγωνισμός στο διαδίκτυο, η κοινόχρηστη οικονομία, ζητήματα γεωργίας, αερομεταφορών, ε, διεθνής συνεργασία και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. και βέβαια ο δημοκρατικό Ελληνικός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι. Μια ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού είναι πάντα ένα εργαλείο για να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ και θα ήθελα να ακούσω τα δικά σας τα σχόλια. Αλλά Βεβαίω, όπω είπα, αναμένω τη συνεισφορά σα συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Από το ΕΛΚ, ο Φούβουλβιο Μαρτουτσέλο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στις αρχές του 19ου αιώνα στο Ellis Island υπήρχε μια επιγραφή που έλεγε ε, δεν χρειάζεται, δεν αρκεί το να είναι κανείς Ούγγρος που υπονοούσε ότι έτσι κι αλλιώς ε, θα υποστήσει και άλλους ελέγχους ε, στην Αμερική. Γιατί το λέω αυτό, διότι θέλω να πω ότι όλο αυτό που συζητάμε ε, ξεκίνησε επικοδοματικά. Στην αρχή ήταν ε, η υπερηφάνεια του Ούγκρου εισηγητή που του έδωσε έτσι κάποιον αέρα. Μετά βέβαια αυτό δεν αρκούσε. Όλοι μας συνειδητοποιήσαμε ότι η στρέβλωση του ανταγωνισμού είναι τροχοπέδι για την ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι σημαντικό να αρθούν όλα τα εμπόδια εις βάρος της, ε, του ανταγωνισμού γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν ανταγωνιστικές τιμές και να ε, τηρηθούν, να παραμείνουν στη ζωή όλες αυτές οι επιχειρήσεις που δίνουν ζωή στην αγορά. Πολύ συχνά το κράτος ε, αλλάζει τη νομοθεσία, επηρεάζει τον ανταγωνισμό και εγώ επ' αυτού θέλω να πω όσον αφορά αυτή την έκθεση. Η έκθεση κατευθύνεται προς μια κατάσταση όπου στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ε, και θα πρέπει λοιπόν η Κομισιό να δει τι μπορεί να κάνει για να άρει τα εμπόδια. Από τώρα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάποια θέματα θα πρέπει αναμφίβολα να εξεταστούν περαιτέρω και μετά ε, θα έχουμε την προκατακτική συνεδρίαση του ΕΛΚ που θα δώσει την ε, τελική κατεύθυνση. Εγώ θέλω να σας πω ότι αναγνωρίζω στον εισηγητή ότι έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και ότι έλαβε υπόψη του όλες τις απόψεις ε, που εκφράστηκαν από τους καθηγητές στις δύο αυτές συναντήσεις που είχαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Άντρελόνς από το Ευχαριστώ. Θέλω I do να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πραγματικά με μεγάλη προθυμία θέλησε να συζητήσει και να ε, βρει μεγάλη πλειοψηφία για τις ε, τροπολογίες. Ε, ε, ακόμα όμως δεν έχω πιστεί ότι φέραμε αυτή την υπόθεση σε αίσιο πέρας. Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα θεωρώ ότι η ομάδα μου δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει την έκθεση με τη σημερινή μορφή, αλλά μαθαίνω από τον εισηγητή ότι συνεχίζονται συζητήσεις για ε, το κείμενο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί θα ήταν κρίμα να μην συμφωνήσουμε η εσωτερική αγορά, η πολιτική ανταγωνισμού είναι στην καρδιά και τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάτι που να μπορούν να υποστηρίξουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Καλή τύχη, θα σας στείλω και εγώ μερικές προτάσεις για συμβιβαστικές τροπολογίες. Για την ουσία της έκθεσης τώρα αυτή καθ' αυτή, εστιάζουμε κυρίως σε θέματα ανταγωνισμού και αυτό θα πρέπει να κυριαρχεί στις σκέψεις μας τα φορολογικά που θεωρούνται συγκαλυμμένες κρατικές ενισχύσεις έχουν σημασία στη συζήτησή μας και κατανοώ αυτό που ζητούν ε, πολλές ομάδες να μπει στην έκθεση. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ε, το παρατραβήξουμε και να ζητήσουμε ε, φορολογική ένωση, ολοκλήρωση, κοινή ενοποιημένη βάση φορολογητέα κτλ. για τη φορολόγηση των ε, επιχειρήσεων και σε ό,τι αφορά τα φορολογικά που συνιστούν κρατικές ενισχύσεις η συζήτηση είναι πολύ πιο βαθιά και ουσιαστική θα πρέπει να δούμε πώς το συνδυάζουμε και με την ασφάλεια δικαίου. Αν δείτε ποιες κρατικές ενισχύσεις χρησιμοποιούνται στα κράτη-μέλη, θα ζητηθεί από κάποιες εταιρείες να αποζημιώσουν, να επιστρέψουν κάποιες κρατικές ενισχύσεις. Ε, και πώς θα τα ζητήσουμε αναδρομικά και με τόκους. Έτσι. Χρειάζεται να έχουμε και περισσότερο κόσμο στην πολιτική ανταγωνισμού για να παίρνονται αποφάσεις πιο γρήγορα για την αρμοδιότητα αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, αλλά αυτό νομίζω δεν θα προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, συμφωνούμε απολύτως ε, ε, να είναι ανεξάρτητη η Γενική Διεύθυνση ε, Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στο χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων. Να παραμένουμε εμείς στα γεγονότα και να μην επεμβαίνουμε σε έρευνες κατά τη διάρκεια των ερευνών αυτών. Γενικά ελπίζω να τα βρούμε και να πείσετε και το ΙΣΙΑ να σας υποστηρίξει. Ευχαριστώ. Γκουε. Η Παλώμα Λόπεθ ε, Μπερμέχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή δουλειά του, για τις συμβαστικές τροπολογίες που προτείνει και επίσης ε, δέχτηκε και πολλές από τις δικές μας τροπολογίες. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι η έκθεση αυτή προσεγγίζει ε, τα αιτήματα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουμε περιοριστική θεώρηση του ανταγωνισμού αλλά να είναι ένα μέσο λειτουργίας της αγοράς ε, λαμβάνοντας υπόψη κάποια εξωτερικά δεδομένα. Στη Γεωργία βλέπουμε επιτέλους ε, να ε, λαμβάνεται υπόψη και ευχαριστούμε και πάλι τον εισηγητή μετά από μεγάλες προσπάθειες. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την φοροδιαφυγή. Το κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να κρύβεται, θα πρέπει να λάβει ε, θέση απέναντι στα όσα κάνει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Χαιρόμαστε που εκφράζονται οι ανησυχίες μας για την συγχώνευση Μπάγερ Μονσάντο. Κάτι που μας λείπει είναι η τροπολογία μας 438 για την πρώην Επίτροπο Κρούς. Στην προηγούμενη έκθεση ανταγωνισμού εμείς επικρίναμε αυτό το σύστημα ε, των περιστρεφόμενων θυρών στην ε, ηλεκτρική ενέργεια όπου βολεύονται κάποιοι πρώην αξιωματούχοι. Ε, δεν μπορούμε τώρα σε αυτή την περίπτωση ανταγωνισμού να σιωπήσουμε. Ελπίζουμε κάτι να γίνει με την τροπολογία αυτή. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με την πορεία της έκθεσης και με τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Thank you you. Ευχαριστώ. Πράσινοι απόντες. Άλλος. Η Μπέτρεξ Φων Στόρχ. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Berichterstatter. Κύριε Σιγητά, η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την ετήσια εκτίση για την ε, πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή δημιουργεί ένα πεδίο όπου μπορούν να λειτουργήσουν οι παίκτες της αγοράς, δημιουργεί το πλαίσιο, πρόκειται για ένα φιλελεύθερο στοιχείο που υπάρχει βεβαίως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ σωστά συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά τις ε, τροπολογίες και τις ε, συμβαστικές προτάσεις είμαι ε, λίγο επιφυλακτική. Στην έκθεση αυτή δεν μπορούμε να θίγουμε θέματα τα οποία δεν σχετίζονται με την πολιτική ανταγωνισμού. Παρακαλώ η έκθεση να είναι συνοπτική, να στοχεύει σε πολιτική ανταγωνισμού και να μην είναι ευκταϊπότη για όλα τα φορολογικά θέματα για κοινή φορολογική βάση και για οτιδήποτε άλλο, γιατί σε τελική ανάλυση η φορολογική πολιτική είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, όσον αφορά την ε, πολιτικής συνοχής αλλά και πάρα πολλά άλλα θέματα. Αυτά είναι θέματα που δεν έχουν καμία σχέση και καμία θέση στην έκθεση περί πολιτικής ανταγωνισμού. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας και τον φίλο Τίμπορ Σάνι με εκπλήσει πάρα πολύ αυτό που είπε η προλαλήσασα, λέγοντας ότι η φορολογική πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι αγνοείς όλα αυτά που έχουν γίνει εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θυμάμαι μια ομάδα εργασία που είχε συσταθεί πριν από 10 χρόνια κάτι τέτοιο υπό την κυρία Πριμαρόλο που είχε στόχο ακριβώς να εξετάσει θέματα ανταγωνισμού από την φορολογική σκοπιά. Άρα Υπάρχει σχέση για το πώς επηρέαζε αρνητικά η φορολογία τον ανταγωνισμό και δεν είναι τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενεύει σε θέματα φορολογικά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Ελπίζω οι συμβασμοί να μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε αυτή τη στρατηγική που είναι πάρα πολύ αποτελεσματική για να προχωρήσουμε ε, για τον ελεύθερο και θεμητό ανταγωνισμό και μη ε, ε, στρεβλωμένο μάλλον. Ευχαριστώ, εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις αυτές νομίζω παρουσίασαν αρκετά καλά τον πυρήνα της δουλειάς που κάνουμε τώρα και είναι νομίζω ένα μήνυμα προς το ΕΣΥΑΡ και είμαι και εγώ αρκετά αισιόδοξο όπως και εσείς ότι στις επομενες δυο δύο-τρεις ωρίτσες θα επιτύχουμε όλους τους ε, στόχους, ε, τους συμβαστικούς που έχουμε. Κατόπιν και προσκαλώ τους ε, συναδέλφους των διαφόρων ομάδων να δώσουν το εξής μήνυμα. Όποιος θεωρεί ότι κάποιες τροπολογίες του δεν υπάρχουν στην έκθεση, ε, πείτε μου το, σας παρακαλώ, γιατί υπάρχει πάντα η δυνατότητα τελευταία στιγμή να κάνουμε κάτι για να περιλάβουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν ε, είναι στην έκθεση. Και ξανά πρέπει να ξεκαθαρίσω το εξή. Εγώ ως συγητής θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι να συνοψίσω τις δικές σας απόψεις, συνάδελφοι. Οπότε, εάν σε κάποιο τομέα, όπως φορολογία, έχω 50 προτάσεις, ε, δεν μπορώ να πω είναι πολλές ή λίγες. Έτσι ε, το βλέπει το Κοινοβούλιο. Και η έκθεση αυτή πρέπει να δει τις ε, τρέχουσες απόψεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το όπως είπε η κυρία Μπερίστα, τα πράγματα αλλάζουν. Πριν από 10 χρόνια είχαμε μια άλλη έκθεση. Σε 10 χρόνια από σήμερα έχουμε πάλι μια διαφορετική έκθεση. Είναι ένα θέμα που αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες και τους εκπροσώπους βεβαίω των πολιτών. Και έτσι κάθε μέρα ακριβώς δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες της ε, εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι η λέξη κλειδί. Και προφανώς ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι στην έκθεση αυτή αντικατοπτρίζονται τα συμφέροντα των πολιτών. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και ελπίζω τις επόμενες μέρες ε, να επιτύχουμε πρόβλημα. Και αν έχω ξεχάσει κάτι, όπως είπα, η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε αυτή την πρόοδο. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε το Φλεβάρι στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λήξη συνεδρίασης. Επόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα, 5 του μηνός Δεκεμβρίου, 3 με 6.30. Πρέπει να σας ανακοινώσω και να σας θυμίσω ότι έχουμε κοινή συνεδρίαση 1η Σεπτεμβρίου με τη ΛΥΜΠΕ την 5η 8 με 9 το πρωί μεθαύριο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος.